Λοιπόν, παρακαλώ, ησυχία. Αρχίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω Ιταλικά, λέει η Πρόεδρος. Καθίστε όμως πρώτα, για να αρχίσουμε. Ωραία. Σας καλωσορίζω όλους. Σήμερα το πρωί Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωινό γιατί θα ψηφίσουμε επί σημαντικών θεμάτων όπως την ψηφιακή ενιαία αγορά και χαίρομαι διότι σήμερα μπορούμε να εγκρίνουμε μία έκθεση της κυρίας Κάμερβέρτ που είναι πολύ σημαντική για την στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά που αφορά πολλές επιτροπές, αλλά εμείς έχουμε τον ουσιώδη ρόλο. Αργότερα θα μας παρουσιαστεί και μία έρευνα σε σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε αντιρρήσεις επί σημερινή ημερήσιας διάταξη, αν όχι προχωράμε το δεύτερο θέμα, ε, δεν ξέρω κατά πόσο είδατε τα πρακτικά της 15ης Οκτωβρίου, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεχίζουμε. Και ε, ως προς τη διερμηνία έχουμε Ιταλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, ε, Αγγλικά, ε, Ελληνικά, Ουγγρικά, Εστονικά, Σλοβενικά, Δανέζικα, Λετονικά και Μαλτέζικα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή και ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε αποστείλει ένα υπόμνημα για το, για, την, για το βραβείο Λουξ που ξέρετε ότι είναι το μεγάλο βραβείο για στην ε, ευρωπαϊκή κινηματογραφία έχουμε τρία έργα, πολύ όριμα έργα και που παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον. Χτες είχαμε μία παράλληλη προβολή δύο από τα ε, τρία έργα σε πολλές ε, ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι οι περίφημες Lux Days και ήταν κατάμεστες οι αίθουσες. Παρουσιάστηκε πρώτα το Mustang και μετά το Mediterranean. Δέκα χώρες συμμετείχαν με κινηματογραφικές ε, αντίστοιχες αίθουσες. Ήταν ένα ευρωπαϊκό γεγονός και θα αποδοθεί και το βραβείο. Μέχρι τις 23 ε, Νοεμβρίου μπορείτε να ψηφίσετε, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, γιατί ο βραβευτής ορίζεται από εμάς τους ευρωβουλευτές. Έχετε όλες ε, τις λεπτομέρειες για τις προβολές εντός κοινοβουλίου σε πολλές χώρες όπως και τη δική μου, σε συγκεκριμένα φεστιβάλ Συμμετείχαν ε, οι τρεις ε, φιναλίστ γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ε, βοηθήσουμε να γίνει γνωστή αυτή η εμπειρία. Όπως ξέρετε, το βραβείο θα αποδοθεί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου υπό την Προεδρία του Προέδρου Σούλτς. Και θα είναι παρόντες και οι τρεις φιναλίστικες. Όπως ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει υποτιτλισμό σε 23 ε, γλώσσες, γιατί σημαίνει ότι θα διαδοθεί εντός και εκτός Ευρώπης. Όλα βέβαια τα έργα. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, συμμετάσχετε όλοι στην ψηφοφορία. Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω και κάτι άλλο. Στις 3 ε, Δεκεμβρίου θα γίνει μία διάσκεψη διακοινοβουλευτική που προωθεί η Επιτροπή Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και ε, Νεότητας με τα 28 Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, από όσο ξέρω, υπάρχουν τουλάχιστον 14 ε, πρόεδροι επιτροπών που θα είναι παρόντες και θα εκπροσωπηθούν και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλή ισορροπία και ως προς το θέμα της, ε, της εκπαίδευσης και, της, ε, ε, και των νέων και όπως ξέρετε και ο Επίτροπος προωθεί αυτό το θέμα γιατί δεν θέλω να μιλάμε για τους νέους αλλά με τους νέους. Το Youth Forum λοιπόν αφορά τις τέσσερις αρχικές ομιλίες και ένας νέος θα είναι σε κάθε πάνελ. Έχουμε τρία πάνελ και θα γίνει λόγος και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε καλέσει και τον εκπρόσωπο της ΕΤΕ που θα μας ε, μιλήσει για τις επενδύσεις μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων για τους ε, νέους και την εκπαίδευση. Ελπίζω να είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, και τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη να είναι παρόντα γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον μας γιατί μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια για να αναγνωρίσουν και την εργασία της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω Επίσης, Α, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Κάτι που συμμερίζονται αρκετοί συνάδελφοι. Όπως ξέρετε, μας απεστάλλει... Με συγχωρείτε, αποστήλαμε μία επιστολή στον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς για ένα θέμα το οποίο θίξαμε άτυπα που έχει ως εξής. Θα θέλαμε και εμείς και το Συμβούλιο στα τέλη Δεκεμβρίου να ασχοληθεί με το θέμα, δηλαδή το 2018 να κηρυχθεί έτος ευρωπαϊκής κληρονομιάς η Ευρώπα Νόστρα και άλλοι οργανισμοί και φορείς, πολιτισμικοί φορείς, έθιξαν το θέμα και μιλήσαμε για την ανησυχία μας, διότι θα πρέπει ε, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε και τα θεματικά έτη, ευρωπαϊκά έτη. Κάτι το οποίο τίνει να καταργηθεί. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του μας, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό συμμερίζονται και οι επικεφαλής αντιπροσωπιών στους συντονιστές και ασχοληθήκαμε και, με, και μεθά μετά της υπό την κυρία Μογκερίνη. Το θέμα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι πιο παρόν ως δικαίωμα για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο και με κατεπίγουσα βοήθεια τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δηλαδή να προβλέψουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και στους προσφυγικούς καταβλισμούς σε τρίτες χώρες. Αυτό θα μας απασχολήσει και μελλοντικά γιατί στο Στρασβούργο θα υπάρξει μία πρόταση ψηφίσματος που προβάλλει η Επιτροπή Ανάπτυξης. Σταματώ εδώ και τώρα περνάμε άμεσα στην γνωμοδότηση που πρέπει να ψηφίσουμε για μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά της κυρίας Κάμερβερτ. Σας υπενθυμίζω ότι στις 9 Ιουλίου η διάσκεψη των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η Ήτρε και η ΙΜΚΟ είναι οι αρμόδιες επιτροπές σε δυνάμει του άρθρου 55, αλλά ζητήσαμε εμείς και η ΕΜΠΛ, ΚΟΥΛΤ, Γιούρι και ΛΥΜΠΕ να συνδεθούν δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία γνωμοδότηση, με, μία ενισχυμένη γνωμοδότηση. Η κυρία Κάμερβερτ ε, παρουσίασε το σχέδιο 21 Σεπτεμβρίου. Είχαμε 183 τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία με τους ε, σκιώδεις. Έφτασε λοιπόν σε ένα κείμενο με βασικούς συμβασμούς που είναι πολύ καλά εξισορροπημένο. Πριν, το, πριν περάσουμε στην ε, ψηφοφορία θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε την κάρτα σας και αν η Πέτρα θέλει να πει δύο λόγια πριν από την ε, έναρξη της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο το έργο που είχαμε να εκτελέσουμε Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές, αλλά και τη γραμματεία της Επιτροπής, αλλά και των πολιτικών ομάδων. Όλοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε έτσι ώστε να ε, καταφέρουμε να δημιουργήσουμε στο δυνατόν περισσότερους συμβιβασμούς και να ταξινομήσουμε ε, τα πράγματα ανάλογα με την ε, απλότητα ή την σημασία που είχαν. Καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε με, τους, ε, με τη συνεργασία αυτή σε μια γνωμοδότηση που ε, πιστεύω θα ικανοποιήσει τους περισσότερους. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο έργο και γι' αυτό θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν γι' αυτό. Οι συμβιβασμοί σίγουρα δεν ήταν κάτι το εύκολο, δεν καταφέραμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, όμως ελπίζω ε, στο τέλος να καταφέρουμε να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία για αυτήν την τόσο σημαντική έκθεση η οποία αναφέρεται στη μεταρρύθμιση της οδηγίας 2010 κάθετος 13. Εμείς ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού είμαστε η αρμόδια επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν με την έκθεση αυτή πιστεύω πως θα στείλουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το ποια κατεύθυνση ε, πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πέτρα. Ευχαριστώ και τη γραμματεία για τη σημαντική της ε, εργασία και βεβαίως και τους σκιώδεις και αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, κατά πόσο να έχουμε ονομαστική, τελική ονομαστική ψηφοφορία. Νομίζω ότι έτσι προβλέπεται. Ωραία, εντάξει. Δεν είναι κάτι το ασύνηθες. Περνάμε στον πρώτο συμβιβασμό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Με συγχωρείτε, για τον 2 ε, θα γίνει ε, ονομαστική, όπως και στην τελική. Για να ζητηθεί ονομαστική, δυνάμει του άρθρου 208 του κανονισμού, θα πρέπει το 1 τέταρτο των μελών να εκφραστούν υπέρ στην ε, περίπτωσή μας τουλάχιστον 8 βουλευτές. Εάν ε, συμφωνείτε, θα ήθελα να το εκφράσετε τώρα, γιατί δεν προβλεπόταν. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Λοιπόν, ποιοι θέλουν την ονομαστική, μόνο τρεις τάσσονται υπέρ, τέσσερις, Ωραία. Ξανά, ποιοι θέλουν ονομαστική. Τρεις συνάδελφοι, ποιοι τάσσονται κατά. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται καν. Λοιπόν, συμβιβασμός 2, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3, εκ νέου υπάρχει αίτημα ονομαστικής. μπορούμε να κάνουμε ένα πακέτο, να τα δούμε on block. Εάν συμφωνείτε, μια για πάντα υπέρ της ονομαστικής για, όλες, για όλους τους συμβασμούς, τότε θα γίνει ονομαστική. Ποιοι τάσσονται υπέρ της ονομαστικής για όλους τους συμβιβασμούς. Δύο. Τρεις. Άρα δεν υπάρχει πλειοψηφία και άρα δεν υπάρχει ονομαστική για κανένα συμβασμό. Τρία. Συμβασμός τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβασμός. Με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 50. Υπαριθμό 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές Συγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. 5. Με συγχωρείτε, δεν έχω τα γυαλιά μου. Δεν έχω τα σωστά γυαλιά. Λοιπόν, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά, υπέρ, ξανά σας παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπορούμε να ελέγξουμε αν το επιθυμείτε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 57. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 60. Έτσι δεν είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Συμβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8, συμβασμός 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, προφορική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, προφορική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Τον Σύμβασμο 10 εντάξει. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της ε, συμβιβαστικής τροπολογίας 10. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. 76. Υπέρ. Κατά. Υπέρ πάλι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ίσως απορρίπτεται. Ίσως, ίσως. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. Λοιπόν, 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβάσμος 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ίσως απορρίπτεται πρέπει να ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. 70-70. απορρίπτεται. Πέρας. Ναι, ναι, ναι, είναι απόλυτα σαφές. Εγώ έκανα λάθος. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14, σύμβασμος 14 στην επόμενη σελίδα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 16 στην επόμενη σελίδα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 17 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 150 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές ίσως απορρίπτεται αλλά θέλω να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. Απορρέπτεται. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, έκανα εγώ λάθος. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 23 υπέρ. Κατά αποχές, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. δύο υπέρ. Έχω δίκιο, ναι, 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 148. Μίκελς. Πέρας. Εγκρίνεται. 158. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές σας ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται κατά μία ψήφο για μία ψήφο 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία 169 επαληθεύουμε Με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος 170 είναι Πέρας εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 25. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 26. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 27 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, και τώρα τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 3 αποχές. Να συγχαρούμε την Πέτρα, την εισηγήτριά μας. Η Πέτρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτό το ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Και θα ήθελα εδώ να αδράξω την ευκαιρία. Παρακαλώ ησυχία, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν όπως είπα, να δράξω την ευκαιρία όχι μόνο να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συνεργάτες, τους ευρωβουλευτές τη Γραμματεία και τη Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων, αλλά θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες εκφαριστίες μου στην σύμβουλο της ομάδας μας, την κυρία Κοσόβα. η οποία θα εγκαταλείψει την Επιτροπή μας και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Επιτροπή Απασχόλησης. Και πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να την ευχαριστήσουμε για την πραγματικά εξαιρετική συνεργασία και μεταξύ μας και μεταξύ των συναδέλφων από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. της εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον της στην Επιτροπή Απασχόλησης και να πούμε πόσο λυπάμαι που μας φεύγετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θα ήθελα να την ευχαριστήσω διότι ήταν άνθρωπος ιδιαίτερα συνεργατικός και είχε μεγάλες και υψηλές ικανότητες, συνεργάστηκε πολύ καλά με τους άλλους policy advisors και την ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, λέει πρόεδρος και διακόπτη, ναι, Γιώργος. Τώρα στο πρώτο μέρος ε, για το βραβείο Λουξ, στο οποίο δίνεται μεγάλη έφαση. Εχθές όμως, την ώρα της ψηφοφορίας, ήταν η επίσημη παρουσίαση του βραβείου. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Δεύτερο, νομίζω ότι με την ψηφοφορία της σημερινή για το Single Digital Act ε, είναι μια ουσιώδης πρόοδος και θέλω να συγχαρώ την Πέτρα για την ικανότητά της να πω μόνο ότι από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να σας πω ότι ε, α, 7.30 ε, έγινε αυτή η παρουσίαση και η προβολή της, ε, του έργου Μεντιτεράνεα. Θα έπρεπε να έχουμε και τον κύριο Ταγιάννη μαζί μας. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε, διότι ε, αναμεταδόθηκε απευθείας σε όλες τις χώρες. Ε, άρα η κυρία Ροσέτη, όπως ξέρετε, έκανε μια πολύ καλή παρέμβαση, αλλά εμείς μπορούμε ε, σίγουρα να το δούμε και στις πόλεις μας και στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι που ε, εξαρτάται από μας ως προς την ε, νέα ψηφιακή αγορά. Είναι μακρά η πορεία, αλλά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ε, φτάσουμε στους απότερους στόχους. Τώρα έχουμε τρεις εκθέσεις, καταρχήν του κυρίου Ντράγκητσι για την έκθεση «Μαθαίνοντας το σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση» Ξέρετε ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας, σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας έγινε μία ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το θέμα έχει μεγάλη απήχηση γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τις ρίζες μας μέσα στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής ηθαγένειας και είναι ένα θέμα που ε, απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους. Στις 11 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία και στις 19 ε, ε, Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Ντράγκητς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω σύντομα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για το μαθαίνοντας στο σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας πω ποια είναι τα κύρια σημεία και μηνύματα. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, ήμουν απεπισμένος ότι μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο είναι κάτι αναγκαίο στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βρισκόμαστε, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης έχουν τις επιπτώσεις τους τα τελευταία χρόνια. Έτσι οι άνθρωποι αμφισβητούν και τα θεσμικά όργανα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμφισβητούν την ίδια την ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όμως οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της και έτσι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και εντοπίζουν όλο και περισσότερο δημοκρατικό έλλειμμα στις αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φάνηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογέ, όπου μόνο 42,6% των Ευρωπαίων πολιτών και μόνο 27,8% στις ηλικίες 18 με 25 ψήφισαν. Ήταν η χαμηλότερη συμμετοχή από το 1979. Η κατάσταση αυτή μπορεί να διορθωθεί αν ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες και αν ενδιαφερθούν και πάλι για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης. Ο καλύτερος τρόπος είναι η διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περάσει στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να καταλάβουν όταν ανήκουν στην Ευρώπη. Να υπάρχει αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της πολυπολιτισμικότητας Οπότε έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο. Θέλω εδώ να τονίσω τη σημασία που έχει και την ανάγκη που βλέπω εγώ για την ευρωπαϊκή διάσταση στο σχολικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο έχει αγνοηθεί για χρόνια. Το 1976 ξεκίνησε μια πρώτη δράση στον τομέα αυτό. Η ευρωπαϊκή διάσταση λοιπόν συνεχώς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Όμως η διάσταση αυτή είναι περίπλοκη και πολυεπίπεδη. Γι' αυτό και η έκθεσή μου επικεντρώνεται σε ένα στοιχείο μόνο, που είναι μαθαίνοντας το σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή διάσταση δηλαδή στην εκπαίδευση. Και η επιλογή αυτή ξεκινάει από το γεγονός ότι οι νέοι πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες καλούνται να γίνουν αργοί πολίτες μέσα σε, ένα, σε μια παγκοσμιοποίηση και σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο. Γι' αυτό χρειάζονται στέρεες βάσεις και γνώσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να έχουν άποψη για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και για τις αξίες στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στη συνέχεια να μπορούν να πειράσουν τις χώρες τους και τις δραστηριότητές τους. Η ιδέα λοιπόν μιας νέας ε, διάστασης ε, στην εκπαίδευση έχει δύο βασικές αλλά αλληλένδετες πτυχές. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά την ίδια τη γεωγραφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία τη και τον πολιτισμό τη και σχετικά με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώ λειτουργούν τα θεσμικά τη όργανα. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με την ε, παραδοχή και νομιμότητα κάθε δημοκρατικού πολιτικού συστήματο που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και μπορεί να νοηθεί με την ευρεία έννοια. Αυτή η διάσταση λοιπόν στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα οι νέοι να μπορούν να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιοτεχνίες που τους χρειάζονται για να μπορέσουν στη συνέχεια να συμμετέχουν σε δημοκρατικές κοινωνίες και να ακουστεί η φωνή τους. Ακόμα και αν η πλειοψηφία των χωρών μελών σιγά σιγά έχει συμπεριλάβει την ευρωπαϊκή διάσταση στο σχολικό πρόγραμμα και στη διδασκαλία, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα με τα ίδια τα βιβλία και τα κείμενα τα οποία μελετούν οι μαθητές. Αν λάβουμε υπόψη μας την περιορισμένη γνώση που έχουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει υλικό σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε μορφή εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Η ψηφιακή κατάρτιση επίσης χρειάζεται περισσότερη προσοχή ώστε να μπορέσει να διδαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες της και στη θεωρία και στην πράξη. Τα βιβλία πρέπει να καλύπτουν περισσότερο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις ηλικιακέ ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μέθοδοι διδασκαλίας στο σχολείο επίσης μπορούν να βελτιωθούν. Είναι ευθύνη και των ίδιων των μαθητών να συμμετέχουν να αντιληφθούν καλύτερα πώς επηρεάζει η Ευρώπη την καθημερινή του ζωή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι δυνατότητε προσφέρονται από τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη εκπαίδευση και του πολιτισμού. Πρέπει αυτά να αξιοποιηθούν πλήρω με σκοπό να προωθηθούν και οι γλωσσικέ δεξιότητε, η ενεργό συμμετοχή στα κοινά, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση και η διαπολιτισμική κατανόηση. Γι' αυτό στην έκθεσή μου υπογραμμίζω την ανάγκη να συνεχίσει η οικονομική στήριξη και να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε δυνατότητες κινητικότητας. Τα προγράμματα αυτά και ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ακόμα περισσότερο να ενημερωθούν όλοι οι φορείς για τις δυνατότητες χρηματοδότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσω τέτοιων προγραμμάτων. Επιπλέον υπάρχουν και πλατφόρμες όπως είναι το Twinning, όπως είναι η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης και το e-Pail για την εκπαίδευση των ανηλίκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, καθώς και αγωγή του πολίτη. Επίσης υπάρχουν και διάφορα δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που προάγουν τη δασκαλία σε θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να προωθούν ακόμα περισσότερο, καθώ επίση και ανταλλαγές μεταξύ αυτών των δικτύων. Τέλο, σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση συστήνει στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να μεριμνούν για τη διαρκή καταλληλότητα των προγραμμάτων σπουδών και των συστημάτων εκπαίδευση, μπαλωμένη και τη επαγγελματική ε, εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου οι συμμετέχοντε να αποκτήσουν τι ικανότητε και δεξιότητε που χρειάζονται μέσα στι σημερινέ ταχύτατα εξελισσόμενε και αλληλοσυνδεδόμενε κοινωνίε. Τα εκπαιδευτικά αιτήματα αντικατοπτρίζουν τι πολύπλοκε κοινωνίε οι οποίε ζούμε και αντιπροσωπεύουν κοινότητε ατόμων με διαφορετική προέλευση που ζουν και μαθαίνουν μαζί. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν παρατέρω δράση για να προωθήσουν στη δακτική ύλη των σχολείων και των πανεπιστημίων τις πολυπολιτισμικές μας αξίες και τις έννοιες του πολίτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμού. Οι αξίες αυτές πρέπει να εμποτίσουν τα προγράμματα σπουδών με οριζόντιο τρόπο. Μόνο έτσι οι ικανότητε των πολιτών θα προωθηθούν και θα μπορέσουν να συμμετέχουν καλύτερα. Τέλος, πρέπει να αναγνωρίσουμε τέτοιε αρμοδιότητες και να υπάρξουν πιο στενοί δεσμοί ανάμεσα στην άτυπη και την επίσημη εκπαίδευση. Τέλος, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να διευκολύνουν τον ρόλο που παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Αυτές είναι κύριες ιδέες που συμπεριλαμβάνω στην έκθεσή μου, που επικεντρώνεται στην ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, συστήνοντας ε, συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ επίσης και για τη συνεργασία σας. Ε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε ε, Ντράγκητσι και συγχαρητήρια για το κείμενο που έχει μεγάλο βαθμό πληρότητας. Θα δώσουμε το λόγο στους Κιώδης και μετά στους άλλους συναδέλφους. Εκτός από τους κιόδης ε, έχουμε άλλους ομιλητές γιατί έχουμε 12 με 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Σουντρόβα. Στέρ, Μάλινοφ, άλλοι, εντάξει. Μάλινοφ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε και πάρα πολύ, αλλά θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να σας εκθέσω την προσέγγιση μου σε σκιώδη εισηγητής. Δεν έχουμε πάντα την ευκαιρία να το κάνουμε, όμως τώρα θα... Ε, ήθελα να πω πως ε, διοργανώνουμε ένα σεμινάριο για τους ε, δασκάλους, του εκπαιδευτικού στη χώρα μου. Τώρα σχετικά με, την, με τις ετροπολογίες θα ε, τις δείτε και μόνοι σας. Θα ήθελα απλά να πω πως ε, θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμβάλλουν πάρα πολύ σημαντικά. Και πιστεύω πως ε, η συνεισφορά τους είναι σημαντική όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, στο έγγραφο αναφέρεται η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος των κρατών μελών την πρώτη κατηγορία, την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας, της διδακτέας ύλη. Εγώ πιστεύω πως ίσως είναι δύσκολο να συμπεριληφθεί στην έκθεση Μένα αλλά ίσως μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι για ορισμένες χώρες Η ιστορία της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο τρόπος μάλιστα που διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας είναι ε, κάτι που μπορεί είτε να εμποδίσει είτε να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιδέα. Και έχουν γίνει κάποιες προτάσεις που βρίσκονται ακόμα σε θεωρητικό στάδιο, αλλά έχει γίνει μια πρόταση σχετικά με το πώς πρέπει να διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να λησμονούμε την ιστορία μας. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ε, τώρα όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις ε, και εκεί. Χρειάζονται καταρχάς εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν όρεξη για να διδάξουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλή οργάνωση από διοικητική πλευράς. Και επίσης θα ήθελα εδώ να πω ότι η υπερβολική πληροφόρηση είναι το ίδιο ε, επιζήμια όσο και η ανεπαρκής πληροφόρηση. Επίσης πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της αρμόδιας ε, αρχής. Οι αρμόδιες αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικέ και για την ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών στην εκπαίδευση. Να αναγνωρίσουμε επίσης τις ε, διαφορές που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα και να προσπαθήσουμε να τις συνδυάσουμε αξιολογώντας ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητα. Επίσης, έχω κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις στις ε, τροπολογίες μου. Για παράδειγμα, ε, υπάρχει μια πρόταση για μια πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική ακαδημία, παιδαγωγική ακαδημία και εδώ θα μπορούσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες στην οργάνωση αυτής της ακαδημίας. Και πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια Ευρωπαϊκή Παιδαγωγική Ακαδημία. Τώρα, όσον αφορά την ε, προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ε, πιστεύω πως πρέπει να σταθούμε στο... στην κατάρτιση των ε, εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία για τα ευρωπαϊκά ζητήματα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι από τα πανεπιστήμια. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υπηρεσία ε, περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν ευρωπαϊκά ζητήματα. Επίσης, πιστεύω πως δεν χρειάζεται να υπάρχουν περιορισμοί στις, ε, στον κλάδο σπουδών για να μπορέσει κάποιος να διδάξει ευρωπαϊκή ιστορία και ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να προέρχεται από το χώρο της ε, φιλολογίας ή των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά θα μπορούσε να έχει σπουδάσει, για παράδειγμα, βιολογία και το ενδιαφέρον του να τον κάνει πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Τώρα, Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε προορατικοί και δεν χρειάζεται να περιμένουμε ε, πολύ. Είναι πιστεύω μεγάλο πλεονέκτημα να αρχίζει η διδασκαλία των ευρωπαϊκών ε, θεμάτων από πολύ νωρίς, από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και θα μπορούσαμε να επιμείνουμε ίσως σε αυτό. Και επίσης ε, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη δασκαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις υποψήφιες χώρες. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Εξαιρετική παρέμβαση, αλλά θα ήθελα να είσαστε πιο σύντομοι, γιατί στις 11 έχουμε την έρευνα. Σέντροβα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Είναι πολύ ωραίο που μπορώ να συνεχίσω κι εγώ τώρα μετά από τον κύριο Μαλίβα γιατί τα σχόλιά του ήταν πολύ επικοδομητικά και πολύ σημαντικά, βρίσκω. Πώς αρχίζουμε να μαθαίνουμε στα σχολεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η εντυπώσεις που έχουμε από τα σχολεία είναι ότι τελικά η Ευρώπη δεν διδάσκεται αρκετά. Ενώ υπάρχουν ευκαιρίες. Τα σχολεία όμως έχουν τόσα άλλα πράγματα, τόσε άλλε υποχρεώσει, τόσα πράγματα να μάθουν στα παιδιά που αυτό το παραβλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον και να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα περνάνε καλά. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτά που είπε ο προλαλής σας. Και αν βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, θα έχουμε συνεισφέρει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή που αναφέρει όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αν προσθέσουμε και αυτή την πρόταση που έκανα εγώ, πιστεύω ότι έτσι εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο η έκθεση και γίνεται πλήρης. Αν έχω κάτι να πω, να επικρίνω, είναι για το σημείο 8 το οποίο αναφέρεται στη δημοκρατική διαχείριση και μεγαλύτερη χρήση της δημοκρατικής ε, διαχείρισης. Η δημοκρατία και ο επαγγελματισμό πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε περισσότερο για τη συμμετοχή των μαθητών και των δασκάλων και όχι να μιλάμε για την άμεση συμμετοχή στην ε, διαχείριση του σχολείου. Μάουρα. Α, δεν ζητήθηκε ο λόγος, με συγχωρείτε. Μαουρ. Για τελευταία φορά σας απευθύνω το λόγο μέλος αυτής της Επιτροπής, διότι παρετήθηκα από Ευρωβουλευτής από τις 25 Νοεμβρίου για να συμμετάσχω στις εθνικές εκλογές στην Ισπανία σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα μου, αλλά ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ισπανική πολιτική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και όλους ε, που συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή, τους βοηθούς, το προσωπικό για την εργασία κατά τον 1,5 αυτό χρόνο, μόλις 1,5 χρόνο συνεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, το οποίο θα πρέπει να, κάτι που θα πρέπει να προωθήσουμε στους, στα θεσμικά όργανα, κάτι που θα το κάνω από τη δική μου πλευρά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξαγάγουμε το προϊόν μας προς τα έξω στις ε, χώρες που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς την ε, εκμάθηση θεμάτων που άπτονται της Ευρώπης ε, στα σχολεία, είναι ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει πάντα. Το ε, έχουμε ενσωματώσει στο πολιτικό μας πρόγραμμα, στο πρόγραμμα του κόμματός μας και θα προωθήσουμε αυτή την έκθεση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομοθετικό ε, κείμενο που να ορίζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Η Ευρώπη είναι ένα σχέδιο των κρατών και όχι τόσο των πολιτών. Άρα κάτι τέτοιο δεν θα σταθεί δυνατόν εάν δεν καταρτήσουμε μια Ευρώπη των πολιτών. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μου γενιά που φτάνουν αργά σε αυτό το σχέδιο, αλλά μιλώ για τους νέους. Διότι οι νέοι είναι οι πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού. Αύριο θα χρειαστούν μία ομοσπονδιακή Ευρώπη, πολύ περισσότερο από ό,τι ορίζουμε εμείς. Γι' αυτό είναι επιτακτικής ανάγκης να ορίσουμε την ε, ιστορία της Ευρώπης που πολλές φορές ήταν, δεν ήταν καθόλου συμφιλιωτική. Χρειάζεται ε, κριτική σκέψη, διότι αυτό θα αντιτάξει τον ευρωσκεπτικισμό. Στην αιτιολογική σκέψη του, της έκθεσης του Ντράγκητσι ορίζουμε τη, τα προγράμματα εκμάθησης της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορώ να πω ότι στην περίπτωσή μου στην Ισπανία δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Συμφωνώ λοιπόν σε αυτή την εξώθηση των κρατών μελών να επικαιροποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα έτσι ώστε να σχετίζονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, δηλαδή από το δημοτικό μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση καθώς και στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ε, μπορείτε να συνοψίσετε διότι έχετε μακρηγορήσει. Ναι, ναι πρόεδρε. Εάν συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και μπορώ να πω ότι στη χώρα μου έχουμε, είμαστε χαμένοι ιδιαίτερα ως προς το θέμα της θρησκείας και της χρήσης της γλώσσας. Χρειαζόμαστε μία ποιοτική εκπαίδευση έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι, αυτή είναι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι ιδιαίτερα που θα χάσουμε ένα συνάδελφο ο οποίος συμμετείχε τόσο ενεργά στην ε, Επιτροπή και που είχε συνεισφέρει σε όλα τα θέματα διευρύνοντας και την θεώρηση των ε, θεμάτων. Δηλαδή ως προς τον πολιτισμό και την ε, πολιτισμική διπλωματία. Σας ε, εύχομαι να τα καταφέρετε στις νέες σας προκλήσεις και ελπίζω να επιτύχετε στους απότερους στόχους σας. Ελπίζω να σας αντικαταστήσει ε, ένας επάξιος διάδοχος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χουντή. Στον κύριο Χουντή, ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο επειδή είναι η πρώτη φορά που παίρνω το λόγο στην Επιτροπή ως νέο μέλος, βλέπετε άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, θέλω να πω για να γνωριστούμε ότι ήμουν Ευρωβουλευτής τα τελευταία πέντε χρόνια σε άλλες επιτροπές, πιο σκληρές, στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Επιτροπή Εξωτερικών. Μεσολάβησε ένας χρόνος όπου θύτευσα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Υπουργός Εξωτερικών της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς επί ευρωπαϊκών υποθέσεων. Οι εξελίξεις με ξανάφεραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή αντικαθιστώντας τον Μανώλη Γλέζο και θα πάρω το λόγο ως κοιόδης συζητητής στο θέμα που συζητάμε σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπα τα βιογραφικά στοιχεία για να δείτε ότι το θέμα το εκτιμώ πάρα πολύ σοβαρά και η προσπάθεια που κάνει ο συνάδελφος και που κάνουμε όλοι για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η, πρώτη μου παρατήρηση είναι η εξής. Αν σωστά εντοπίζει η έκθεση έχουμε κάποια προβλήματα, προβλήματα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε στο πώς αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προσδοκούν και πώς συμμετέχουν, τότε οφείλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι εδώ καλές οι αλλά κατά τη γνώμη μου οι προτάσεις δεν απαντούν και δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα. Έχουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που τα τελευταία χρόνια δεν μετέχουν στις διαδικασίες, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στη χώρα μου εμφανίστηκε το τελευταίο στις τελευταίες εκλογές το 50% να μην παίρνει μέρος στις εκλογές. Τι πρόβλημα λοιπόν εδώ υπάρχει. Είναι άγνοια. Δεν γνωρίζουν καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα. Ή έχουν απογοητευτεί από τις κυρίαρχες πολιτικές που εισπράττουν στην καθημερινότητά τους. Και η απογοήτευση δεν είναι επί της ουσίας της πολιτικής. Είναι γιατί απογοητεύτηκαν διότι σου λέει συμμετέχοντας και ψηφίζοντας κάτι δεν εφαρμόζεται διότι έρχεται κάτι άλλο και λέει αυτό θα γίνει και δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Επομένως η ενεργοποίηση του πολίτη μοιάζει άχρηστη. Τι τον καλούμε λοιπόν. Για να είμαι κωδικοποιημένος θα κάνω ε, τροπολογίες στο θέμα αυτό. Αν λοιπόν σωστά τοποθετεί το θέμα ότι εκπαίδευση σημαίνει, αυτή η διαδικασία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι γνώση της γεωγραφίας, της ιστορίας, και άλλων στοιχείων που συγκροτούν αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οφείλω να κάνω την παρατήρηση ότι αυτή η γνώση πρέπει να δίνεται σωστά και πλήρω. Με σκοπιμότητα να αναδείξει τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα προσφυλές. Πόσοι γνωρίζουν από πού προέκυψε το θέμα Ευρώπη. Κατά την ελληνική μυθολογία η Ευρώπη ήταν μια βασιλοπούλα της Φινίκης δηλαδή της σημερινής περιοχής του Λιβάνου, το υπογραμμίζω του Λιβάνου, για να έρθουμε στην επικαιρότητα τη σημερινή. Πώς αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό. Επομένως, για να μην επεκταθώ περισσότερο, σωστή γνώση της γεωγραφίας, της ιστορίας, για να μπορέσουν να βγαίνουν και τα μηνύματα που θέλουμε σύμφωνα με τις αξίες που θέλουμε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, η δεύτερη διάσταση είναι εκπαίδευση, αγωγή του πολίτη. Ερώτημα. Πόσοι γνωρίζουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πραγματικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες στο τελευταίο διάστημα ακούνε Dijsselbloem. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Dijsselbloem. Ακούνε Eurogroup. Αυτό αποφασίζει. Μα αυτό δεν είναι θεσμός σύμφωνα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι καταλαβαίνει ο άλλος όσον αφορά τις δικέ του δυνατότητε. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο γιατί θέλω να πω λοιπόν ότι η θεραπεία για μένα το πρώτο σκέλος σωστή και πλήρη ενημέρωση για τη γεωγραφία την ιστορία τις αρχές και τις αξίες που συγκροτήθηκε η ευρώπη και η ευρωπαϊκή ένωση για δε το δεύτερο πραγματική αποτύπωση της σημερινής εικόνας που έχει η ευρωπαϊκή ένωση διότι διαφορετικά θα βάλουμε το, πρόβλημα κάτω από το χαλί άλλα θα διδάσκεται άλλα θα βλέπει στην καθημερινότητά του γεγονός που θα το απομακρύνει από τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σταματώ εδώ γιατί ε, θα καταθέσω τροπολογίες όπως αντιλαμβάνω σε μια σειρά σημεία για να βοηθήσω να φτιάξουμε μια καλή έκθεση. Ε, σας ευχαριστώ και σας ε, καλωσορίζω συνάδελφοι. Ξέρω ότι αντικαθιστάτε τον συνάδελφο Γλέζο, τον οποίο είχαμε εκτιμήσει ιδιαίτερα. Είναι ένας ευπατρίδης στη χώρα του, στη χώρα σας και το γνωρίζουμε. Ε, δύο συναδελφοί έχουν το λόγο, Σβέρ και Γιάκονο, για τρία λεπτά σύνολο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Ντραγκίτσι για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. η Ευρώπη έχει και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν είναι μόνο ένα σύνολο διαφορετικών ε, οντοτήτων και ταυτοτήτων και αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα πρέπει να ενισχυθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ε, στο μάθημα της ιστορίας. Πιστεύω πως ε, η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα στο μάθημα της ιστορίας. Πριν από 25 χρόνια δημιουργήθηκαν πολλά νέα κράτη και άλλαξε λοιπόν η διδακτέα ύλη προς ε, αυτήν την κατεύθυνση, προς την παρουσίαση αυτών των ε, νέων κρατών. Τώρα έχουν αλλάξει και πάλι τα πράγματα και βλέπουμε πως υπάρχει μια στροφή στην ε, παγκοσμιοποίηση και στην πανευρωπαϊκή διάσταση. Πιστεύω πως δεν πρόκειται μόνο ε, μάλλον πως η ιστορία δεν είναι μόνο ε, γνώση, στήρα γνώση, αλλά χρειάζεται και ε, εκπαίδευση και ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές αξίες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έκφανση αυτών των ευρωπαϊκών αξιών. Και θεωρώ πως αυτή η αξία πρέπει να τονίζεται στα βιβλία της ιστορίας. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση και πολιτισμική διάσταση και πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν την ε, πολιτισμική αξία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στον χώρο της εκπαίδευσης η διαδικασία μεταρρυθμίσεων της ε, Μπολόνια είναι μία έκφανση της ευρωπαϊκής ιδέας. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα διδάξουμε στην ε, ιστορία και πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, διότι το, η εκπαίδευση είναι εθνική αρμοδιότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η ευρωπαϊκή διάσταση να επεκταθεί στην, ε, στο χώρο της εκπαίδευσης σιγά σιγά, βήμα βήμα. Επίσης, Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται και εκείνη κατάρτιση έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταδώσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην παιδεία. Διάκονο, Έχουμε και άλλους δύο ομιλητές, αλλά έχουμε άλλες δύο εκθέσεις πριν από την παρουσίαση της έρευνας. Θα ήθελα λοιπόν να είσαστε πολύ σύντομοι, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Κατά την άποψή μου, όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα θα μπορούσαν να θεραπευτούν μόνο από την εκπαίδευση. Είναι το κλειδί της επίλυσης όλων των προβλημάτων που έχουμε και θα έχουμε. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο αυτό το θέμα Αγαπητέ Ντράγκητσι, θα είμαστε κι εμείς ε, δίπλα σας και θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα και μόνο. Θα πρέπει να υπάρχει ενσυνειδητότητα από τους Ευρωπαίους πολίτες ότι κάθε έθνος αποτελεί μία πρόσμιξη πολλών ιστοριών. Δεν υπάρχουν αυτούσιες οντότητες. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες ε, χρόνια εμπόλεμων σειράξεων και κινητοποιήσεων καθώς και κινητικότητας. Και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απότοκη των κρατών. Ακόμα και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Φάρατζ ε, για να στυλιτεύσει τις άλλες είναι πρόσμιξη άλλων γλωσσών. Και τα παιδιά θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, έτσι ώστε όταν μας ρωτούν από πού προερχόμαστε να μπορούμε να πούμε γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ. Λιμπάτσκα, εντάχει παρακαλώ και τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τον προλαλήσατα, τον κύριο Τεκόν, γιατί η καλύτερη πράγματι αντιμετώπιση είναι η καλή εκπαίδευση. Αλλά ακόμα και η καλύτερη θεραπεία, αν δεν εφαρμόζεται σωστά, δεν αποδίδει. Αν εφαρμοστεί λάθος δηλαδή. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επιπλέον μαθήματα στο ήδη φωτομένο σχολικό πρόγραμμα. Θέλουμε μέσα στο ήδη υπάρχον σχολικό πρόγραμμα να προσθέσουμε κάτι για την αγωγή των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι. Θέλουμε να έχουμε υπόψη μας τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Όπως έχουν πει και άλλοι πάντως, πρέπει οι καθηγητές να είναι καλά εκπαιδευμένοι, καταρτισμένοι, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μεταφέρουν αυτή τη γνώση, αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Στάκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ στηρίζω αυτή την έκθεση. Θα τα πω φιλανδικά. Όχι, δεν θα τα πω φιλανδικά. Καλύτερα θα τα πω αγγλικά και θα μπορούσα να τα είχα πει και φιλανδικά. Λοιπόν, για την εκπαίδευση. Θέλω να σας πω ότι έχουν την αρμοδιότητα οι χώρες μέλη. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ένας συντονισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συντονίσει. Σύμφωνοι. Η πραγματική αρμοδιότητα όμως είναι των χωρών μελών. Όταν ερχόμαστε στο θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δύσκολα μπορεί κανείς να δώσει έναν ορισμό. Καλό είναι όμως να μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι περί τίνος πρόκειται. Η Ευρώπη είναι κοινέ αξίες. Αυτό είναι που πρέπει να τονίζουμε κάθε φορά και να υπογραμμίζουμε παντού και πάντα. Για την κοινή μας ιστορία, και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί όντως η κοινή μας ιστορία είναι διαφορετική ανάλογα με το από πού προερχόμαστε. Θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία ήμουν εισηγητή ακριβώ για το θέμα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Και θυμάμαι ότι είχα ακούσει πολλές και διαφορετικές απόψεις για την ευρωπαϊκή μας ιστορία. Πάντως το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη και τους υπουργούς να κάνουν κάτι σε αυτό το τομέα. Την ε, εκπαίδευση δηλαδή για ευρωπαϊκά θέματα. Και είναι δικιά τους αρμοδιότητα, όπως είπα και στην αρχή. Στηρίζω λοιπόν την έκθεση, στηρίζω αυτό που λέτε. Όντως πρέπει να πιέσουμε τις χώρες μέλη για να το κάνουν, να συμπεριλάβουν στη διδακτική ύλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κλείσει, έχει κλείσει η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και μια πολύ καλή βάση εργασίας. Ε, μπορούμε βεβαίως να υποβάλουμε τροπολογίες μέχρι τις... Ρωτάει η Πρόεδρος. Μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι φέτος, μάλλον το 2016, θα θέσουμε το δίλημα του πώς μπορούμε να επεξηγήσουμε τις επιμέρους ιστορίες των χωρών των κρατών της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις δύο διαστάσεις. Τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση του συναδέλφου Μαραγάλ που θα ήθελα να λάβει το λόγο. Πρόκειται για το Erasmus Plus και άλλα εργασία για την πρόθεση της ε, κινητικότητας μέσα στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Η έκθεση αυτή Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες μέχρι τις 24 ε, Νοεμβρίου, ε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και η ΕΜΠΛ συμμετέχει, δυνάμει του άρθρου 54, άρα και οι δύο επιτροπές θα συνδράμουν και θα γνωμοδοτήσουμε στις 11 Ιανουαρίου του 16 ε, Μαραγάλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε από μια γενική ιδέα για να προσεγγίσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να σκεφτούμε την σχέση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα που έχει η Ευρώπη. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτήν τη σύνδεση, σε αυτή τη σχέση. Ποιες είναι οι συνέπειες. Δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και να τροποποιήσουμε σημαντικά τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ξέρουμε πόσο μεγάλη ανεργία έχουμε. Φυσικά δεν είναι η ίδια κατάσταση σε όλες τις ε, περιφέρειες της Ευρώπης, από 0 μέχρι 50% ανάλογα με το που βρισκόμαστε. Όπως επίσης η εγκατάλειψη του σχολείου πριν να το τελειώσει ένας μαθητής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η επαγγελματική κατάρτιση λοιπόν βρίσκεται στο κέντρο της αντίφασης. Της ανεργίας δηλαδή, είναι αιτία για την ανεργία. Και γι' αυτό θα πρέπει τα προγράμματά μας να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η επαγγελματική κατάρτιση όμως είναι αρκετά περίπλοκη και πολλές φορές δεν είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην αγορά εργασίας. Για λόγους που μερικές φορές είναι και ιστορικοί. Πρώτα απ' όλα υπάρχει διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα στην κάθε χώρα και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε καν ένα ευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης εκπαιδευτικών τίτλων ώστε να αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο την εμπειρία και τα διπλώματα. Από την άλλη μεριά όμως, η Ευρώπη μπόρεσε να έχει σαν βασική έννοια την κινητικότητα, που έχει δείξει τα θετικά της. Με το Εράσμους, το Λεωνάρδο, το Εράσμους Συν τώρα, μόνο θετικές εμπειρίες έχουμε από αυτά όσον αφορά την, κινητικότητα. Με την κινητικότητα εξάλλου αποκτάει κανείς και περισσότερες εγκάρσιες ε, γνώσεις και εμπειρίες. Έπειτα, οι μαθητές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα εμπόδια αντικειμενικά, αλλά και όχι μόνο, για την κινητικότητα αυτή πρέπει να αρχίζουν πιο νωρί να μαθαίνουν ξένες γλώσσε, υπάρχουν ε, οικονομικοί και άλλοι λόγοι, γι' αυτό και μιλάμε εδώ πέρα και για την, ε, το καθεστώς του μαθητευόμενου. Έπειτα, δεν είναι κατάλληλα τα προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας στην Ευρώπη. Τα κέντρα μας επαγγελματικής κατάρτισης έχουν διαφορές μεταξύ τους. Τα παραγωγικά μοντέλα στις διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο ένα συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί κι αλλού. Γι' αυτό λοιπόν, με την έκθεσή μου, θέλω να αντιμετωπίσω όλες αυτές τις δυσκολίες που σας ανέφερα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές μας, να τους προετοιμάζουμε καλύτερα για την κινητικότητα, δηλαδή να μαθαίνουν γλώσσες, να τους συνοδεύουν οι δασκάλοι τους κτλ. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ένα πραγματικά πλήρες ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων. Πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε σε καινοτομίες στα προγράμματά μας για την κοινοτικότητα με διάφορα κέντρα και μεσάζοντες που χρειάζονται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο για τις μεγάλες. Η πρότασή μας απευθύνεται βέβαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοείται. Και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πάρει αυτό το μήνυμα. Να δημιουργηθεί ένα πραγματικό λοιπόν Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής ε, Εκπαίδευσης, να ενισχυθεί κινητικότητα, όλοι οι πόροι του Εράσμους ε, συν να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπάρχουν και στοιχεία συντονισμού που χρειάζονται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μεταξύ των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας, για παράδειγμα Έρασμος ΣΥΝ και Κοινωνικό Ταμείο. Ένα λεπτό ακόμα. πρέπει να απευθύνουμε περισσότερους σπόρους στους σκοπούς αυτούς. Σαν μια πραγματική ευρωπαϊκή κυβέρνηση πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, να χρησιμοποιήσουμε όλους τους σπόρους που χρειάζονται να πάνε στα νέα αυτά δίκτυα τα οποία ενισχύουν την επαγγελματική εκπαίδευση. Το βασικό είναι να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεσματική για να αντιμετωπίσουμε και την εγκατάλειψη του σχολείου πρόωρα και την ανεργία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση με τους σκιώδεις εισηγητές με πολύ θετικό πνεύμα και με τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Απασχόλησης ώστε να λάβουμε υπόψη μας και την δικιά τους άποψη. Φυσικά πολλά μπορούν να προσθεθούν εδώ και να αλλάξουν ακόμα, πολλά θα μπορούσατε να επικρίνετε. Εγώ συνόψισα, ίσως πολύ συνθετικά, όπως και να έχει το πράγμα. Αποτελεί μια βάση για να προχωρήσουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω για τις επαφές που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους αρμόδιους εκεί, οι οποίοι μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η κατάσταση. Τους ευχαριστώ ειλικρινά και ελπίζω να συνεχιστεί εξίσου καλά η συνεργασία μας και στο μέλλον. Περιμένω τώρα τις δικές σας τις παρατηρήσεις και σχόλια. Η δουλειά αυτή ελπίζω να μπορέσει να χρησιμεύσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει πιο αποτελεσματική και πραγματική την ε, πολιτική μας για την εκπαίδευση. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο προτάσεις στον ε, προϋπολογισμό και ελπίζω να προχωρήσουν στη διαδικασία. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθούν οι ιδέες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Έχουμε ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες από αυτή την έκθεση γιατί θα αποφανθούμε κι εμείς και στο θέμα της διαβίου μάθησης και της πρόσβασης στο Erasmus Plus όλων με αξιοπρέπεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αναγνωρισιμότητα των βαθμών του Erasmus, Κάτι το οποίο δεν ισχύει αμέσα. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο τώρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με την Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, ποιοι θέλουν το λόγο για να κλείσουμε τον κατάλογο Μωράν Σαρτιέ, Λιμπάτσκα. Καταρχήν, πρώτον ε, η Σκιώδης. Καμερέβερτ και Μόργανο. Λυπάμαι, δεν μπορώ να δεχτώ άλλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την εισήγησή σας που υπογραμμίζει και τη σημασία αυτής της έκθεσης θα πρέπει να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να είμαστε αποδοτικοί γιατί το θέμα είναι ύψης τη σημασίας. Το πρώτο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ γενικότερα έχει ως εξής. Μιλάμε για τον έρασμος ε, συν και την κινητικότητα στην κατάρτιση. Δεν θα πρέπει δηλαδή εδώ να μιλάμε για τον έρασμο ε, γενικά. Το έρασμος πλάς είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, όχι μόνο αυτούς που έχουν κάποιο δίπλωμα, αλλά αυτούς που δεν έχουν επαγγελματικά προσόντα, τους οποίους τα προσφέρουμε, γιατί δεν είχαν αυτή την ευκαιρία από τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου και κύριε Μαραγάλ θα ήθελα να παρέμβω σε ένα από τα σημεία της έκθεσής σας. Εγώ θα ήθελα να αποσαφηνίσω τρεις ιδέες που θα πρέπει να εγγραφούν στην έκθεση. Καταρχήν η κινητικότητα θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των ανισοτήτων. Η πρόσβαση στην κινητικότητα θα πρέπει να είναι ένα διορθωτικό στοιχείο στις ανισότητες που είναι απότοκες της κατάρτισης της ακαδημαϊκής κατάρτισης ε, η οποία οδήγησε στη μαζικοποίηση των διπλωματούχων αλλά όχι στην εξατομίκευση, στην εξατομίκευσή τους τις ανισότητες γεωγραφικού τύπου, τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί είδαμε και στον έρασμο ότι υπήρξαν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που διαγράφονται μέσα στα πλαίσια της πρόσβασης στην κινητικότητα και επίσης ανισότητα μεταξύ αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος. Δηλαδή οι ευκαιρίες κινητικότητας δεν είναι ίδιες. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την πολιτική μας σε αυτή την ε, μείωση των ανισοτήτων. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το εξής. Το θίγει και ο κύριος Μαραγάλ. Είναι τα μέσα κινητικότητας. Εμείς διαθέτουμε τέτοια μέσα, μέσα κινητικότητας. Θα πρέπει όμως να είναι σαφή, προσβάσιμα, κατανοητά και να βάλουμε τους κρίκους αυτής της αλυσίδας σε μία σειρά. Βεβαίως το Erasmus Plus θα πρέπει να σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΚΤ αναλαμβάνει την κινητικότητα ε, εκείνων που δεν διαθέτουν δεξιότητες ή επαγγελματική κατάρτιση για να συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο. Και είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες, επιστροφή στην κατάρτιση. Πρέπει να συνοψίσετε. Το τρίτο θέμα που δεν υπάρχει σε αυτή την έκθεση αφορά τον ε, θελούσιο χαρακτήρα συμμετοχής στον εθελοντισμό. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι ο εθελοντισμός ε, φύγει άλλου άλλες κατηγορίες νέων, εκείνο που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Και οι περισσότεροι εθελοντές που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα προέρχονται από, το, από μη αστικό περιβάλλον, αγορατικό περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα μεγάλο χάσμα. Και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε τρεις βασικές ιδέες την ε, ε, προσωπική κατάρτιση και την απασχολησιμότητα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το ικρίο μας το οποίο θα πρέπει να βασιστούμε έτσι ώστε να έχουμε μία ε, επικοδομητική έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι, διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουν. Τρία λεπτά μάξιμουμ. Λιμπάτσκα, Κάκιμε Καμερέβερτ και Μόργαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη, μια που δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή διότι εντοπίζει με πολύ σωστό τρόπο τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχω περίπου 12 τροπολογίες που θα υποβάλω, οι οποίες τονίζουν κυρίως τις ανισότητες. Διότι υπάρχει από τη μία η... υπάρχουν από τη μία οι κοινωνικές ανισότητες, όπως είπε και η ε, προηγούμενη ομιλήτρια, Και πέρα από αυτό, πέρα από τις ε, ικανότητες, πρέπει να σταθούμε, πιστεύω, και στην προσωπική εξέλιξη του ατόμου. Και να δούμε τι γίνεται με τις ε, υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές για τα προγράμματα Εράσμους στα κράτη-μέλη, οι οποίες λειτουργούν ε, διαφορετικά και από τις οποίες μπορούμε να λύσουμε βέλτιστες πρακτικές. Επίσης... Ε, Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά λόγω οικονομίας χρονού θα είμαι σύντομη. Πρέπει να δοθεί έμφαση στους νέους ανθρώπους στα προγράμματα Εράσμους και Εράσμους ΣΥΝ. Θα μπορούσαν, ε, για παράδειγμα, να ολοκληρώνουν ε, σπουδές και κάποιο είδους επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική ταυτόχρονα. Να υπάρχει δηλαδή ένα ε, διπλό σύστημα εκπαίδευσης που να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και το Erasmus Plus για τους νέους επιχειρηματίες που δεν είναι γνωστό. Κάμε Ρέβερτ, δύο λεπτά. Yeah, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, συνάδελφο κύριο Μαραγκάλ, διότι πιστεύω πως η έκθεσή του είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πιστεύω πως και οι παρατηρήσεις που ακούσαμε από τις ε, δύο συναδέλφους είναι πάρα πολύ σωστές και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ε, έκθεση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε μια πιο πρακτική διάσταση του θέματος. Πριν από λίγες εβδομάδες, δύο-τρεις, ε, οι σοσιαλδημοκράτες διοργάνωσαν ένα συνέδριο που ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα ε, του Εράσμους και Εράσμους ΕΣΥΝ. Είχαμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που αναφέρθηκαν πάρα πολλές ε, πρακτικές λύσεις και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την αναθεώρηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus+. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο αυτά τα προγράμματα, το Erasmus και το Erasmus και όχι μόνο για ε, τους ε, φοιτητέ. Αυτή τη στιγμή το Erasmus είναι συνδεδεμένο με ε, τους ε, φοιτητέ και τους ε, σπουδαστές και δεν χρησιμοποιείται αρκετά μετά η διάσταση και των άλλων προγραμμάτων. Πιστεύω πως επίσης πρέπει τα προγράμματα αυτά να είναι πολύ πιο ευέλικτα και να απλοποιηθεί περισσότερο η διαδικασία οργάνωσής τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Στην Επιτροπή μας ε, στόχος μας είναι να απλουστευτούν όλες οι διαδικασίες, αλλά δυστυχώς βλέπω πως ε, τείνουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Πιστεύω πως ε, θα μπορούσαμε να, και καθήκον μας μάλλον θα ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολύ ε, μικρότερα, πολύ απλούστερα έργα να πραγματοποιηθούν. Αλλά πιστεύω πως Χρειάζεται επίσης και να ξεδιαλέξουμε κάπως ε, τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε, να δούμε ποια είναι πραγματικά χρήσιμα, ποια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και ποια ίσως χρηματοδοτούνται υπερβολικά. Επίσης ε, στο θέμα του προϋπολογισμού πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε καλύτερη ε, κατανομή πόρων για τα πιο ωφέλιμα προγράμματα. Δηλαδή είναι κάποια πρακτικά ζητήματα τα οποία πιστεύω πρέπει να εξετάσουμε, διότι Θεωρώ πως το Erasmus Εσύ είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα και πρέπει να φροντίσουμε αυτή η ιστορία επιτυχίας να ε, συνεχίσει και να μεταφερθεί και σε άλλα προγράμματα και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριλάβουμε περισσότερους νέους αλλά και όχι μόνο στην ε, κινητικότητα στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό όργανο αυτό που έχουμε στα χέρια μας όμως πρέπει να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Τσβέρ και Μόργαν και κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Σύντομος, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ ε, συγχυτή για αυτό το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης. Το Erasmus Plus είναι πραγματικά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Όμως αναρωτιέμαι εάν έχουμε όντως περιπλέξει τα πράγματα. Αν προκαλέσουμε σύγχυση, θα δείξει ε, στο μέλλον τι θα γίνει. Πιστεύω όμως πως έχουμε βελτιώσει την κινητικότητα, δημιουργούμε με το Erasmus είναι καλύτερες προϋποθέσεις, καλύτερη κατάρτιση, καλύτερες δεξιότητες στους νέους ανθρώπους κάτι το οποίο αυξάνει την απασχολησιμότητά τους, έτσι όπως έχει αποδειχθεί στατιστικά. Όμως, τα κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν όσο θα έπρεπε στην ε, διοργάνωση και προώθηση αυτών των προγραμμάτων. Ας ε, μην ξεχνάμε τα προγράμματα της, ε, το πρόγραμμα της Κοπενχάγης. Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Τα κράτη-μέλη, λοιπόν, πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Μόργαν ο τελευταίος ε, ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Μαραγκάλ. Και εγώ εντάχει θα ήθελα να προσθέσω ορισμένες σκέψεις. Η μία είναι μία φιλοδοξία. Θα πρέπει να δούμε τα κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν και να κάνουμε το πραγματικό βήμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πολλές φορές μιλάμε για βελτίωση των επιλογών κινητικότητας για τους νέους. Ή ορίζουμε τις καλύτερες πρακτικές και τις προτείνουμε σε πιλωτικά σχέδια ή διαφορετικά επαναλαμβανόμαστε όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα που αφορούν την αμοιβαιότητα για την κινητικότητα. Και πιστεύω ότι το πρώτο πρόβλημα αφορά μία απλούστευση. Δεν είναι δυνατόν να, επιπλέ, επιπλέκουμε τα θέματα και εάν εξαρτάται από μας θα πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το πέρασμα και θα πρέπει να το κάνουμε ως κοινοβούλιο. Έτσι θα μπορέσουμε ε, τα, ποσά αυτά, με συγχωρείτε, να τα δαπανίσουμε καλύτερα εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, μας απασχολήσουν και άλλα στοιχεία, διότι άλλο η προσφορά εργασίας αλλά όταν δεν υπάρχει εργασία το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί. Το θέμα λοιπόν είναι να ε, γνωρίσουμε καλύτερα το ζήτημα διότι η εγκατάλειψη του σχολείου α, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που διανύουν. Ευχαριστώ συνάδελφε Μόργανο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή θα ήθελε κάτι να μας πει για τη σημαντική αυτή έκθεση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι παίρνουμε το μήνυμα του κύριου Μαραγκάλ που μας ενθαρρύνει να συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε πιο φιλόδοξους ακόμα στόχους στον τομέα της επαγγελματική κατάρτισης. Ιδιαίτερα θέλω να αντιδράσω σε κάποια σημεία. Πράγματι, έχουμε προγράμματα κινητικότητας του Erasmus Συν που λειτουργεί καλά και που μπορούμε μαζί να βελτιώσουμε περισσότερο. Αναφερθήκατε στα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία ότι πρέπει να ανοίξουμε ε, τα προγράμματα αυτά περισσότερο σε ανθρώπους από χώρους που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Επίσης είπατε ότι πρέπει να προετοιμάζουμε τους μαθητές για την κινητικότητα. Έχουμε λοιπόν συστήματα για να τους προετοιμάσουμε καλύτερα, γλωσσικά για παράδειγμα. Αναφερθήκατε επίσης στο ρόλο των ενδιάμεσων και στο ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ενδιάμεσοι αυτοί. Όντως υπάρχουν, είτε είναι οι δήμοι, είτε είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, ε, μας βοηθούν. Θα μπορούσαμε ίσως να αναπτύξουμε και άλλους για να χρησιμεύσουν ακόμα περισσότερο στους νέους. Χωρίς όμως να προσθέτουμε περιτά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά την απλοποίηση, η κυρία Κάμερο Βερτά αναφέρθηκε στην απλοποίηση. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Η γενική μα διευθύντρια, όταν έγινε η ακρόαση πριν από μερικέ εβδομάδε, δεσμεύτηκε προ αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα ανοιχτά, με πολλά έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να βελτιώσουμε ό,τι γίνεται να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Η συγητής θέλει κάτι να προσθέσει εντάχει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ειλικρινά βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή σκέψης, γνωρίζοντας τα μέσα και τις ευκαιρίες και τις εκπληρώσεις στόχων που είχαμε μέχρι τώρα και τα ζητήματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στο ελάχιστο τουλάχιστον. Έχουμε πολλές ε, θετικές εμπειρίες, αλλά δεν μπορούμε να τις γενικεύσουμε. Δεν χρειάζεται να ε, εφευρίσκουμε πολλά πράγματα. Έχουν εφευρεθεί αλλά πρέπει να μαθαίνουμε, να ολοκληρώνουμε και είμαστε πολύ αργοί στην ενσωμάτωση των εμπειριών σε ε, συστήματα. Αυτό σημαίνει πολιτική, αυτό σημαίνει διακυβέρνηση, αυτό σημαίνει ευθύνη των τριών θεσμικών οργάνων. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη της Κομισιό αλλά και των κρατών μελών. Είναι δύσκολο η Επιτροπή να κάνει κάτι παραπάνω από να δώσει μία όθηση προγραμμάτων αν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επικαιροποιήσουν και δεν έχουν τη θέληση να ενσωματώσουν αυτά τα μέσα και να τα απλουστεύσουν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το θέμα του εθελοντισμού τώρα Νομίζω ότι είναι ε, ενδιαφέρον, μπορεί να ενσωματωθεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το εντάξω. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω για ευθύνη κυρίως των ε, δημόσιων θεσμών. Δεν μπορούμε να προσφεύγουμε σε αυτά τα μέσα μόνο. Θα πρέπει να ορίσουμε την δημόσια ευθύνη, τη δημόσια εκπαίδευση, τους οικονομικούς φορείς και θα πρέπει όλα αυτά να μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε αποτελέσματα ως προς την απασχολησιμότητα και την εγκατάλειψη του σχολείου, όπως είπε ο κύριος Μοργάνο. Ως προς την ε, μείωση των ανισοτήτων, όπως ελέγχθη σε πολλές ε, παρεμβάσεις, δεν μπορούμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να συγκλίνουμε την πείρα όλων των ε, περιφερειών. Δηλαδή στη Βάδη Βιρτεμβέργη υπάρχουν άλλοι, άλλα ποσοστά ε, ως προς το δίκτυ ανεργίας των νέων ή στην Καταλωνία όπου ο δείκτης ανεργίας ανέρχεται σε 50% για τους νέους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Μας ε, διέπουν οι ίδιοι κανόνες, αλλά έχουμε αποτύχει σε αυτόν τον τομέα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολλά υποσχόμενη έκθεση. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Υπάρχει το θέμα της συστηματοποίησης. Έχουμε μία πολυεπίπεδη προσέγγιση, εθνική, περιφερειακή, τοπική. Θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα σύστημα. Μιλάμε για Eurochambre, για παράδειγμα. Γιατί να μην μιλάμε για ένα πρόγραμμα πλαίσιο, έτσι ώστε να ε, συγκροτήσουμε καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση. Θεωρώ ότι όπως είπε και η συνάδελφος ε, Καμερέβερτ και έχουμε ε, προβάλει πρόσφατα αφορά το ότι η Επιτροπή μπορεί στους επιμέρους διαγωνισμούς ε, Erasmus Plus να ορίσει αυτά, αυτή τη βαθμολογία η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Θα πρέπει να το κάνει γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Και όπως είπε και η συνάδελφος Μωρέν Σαρτιέ, θα πρέπει να σταθούμε στην άτυπη κατάρτιση. Μην ξεχνάμε ότι στο Erasmus Plus υπάρχει και ο εθελοντισμός και άλλες προσεγγίσεις. Πολύ καλή αυτή η προσέγγιση του κυρίου Μαραγάλ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24 Νοεμβρίου Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Και τώρα περνάμε. Έχουμε 20 λεπτά καθυστέρηση. Να δούμε λοιπόν ε, μία έκθεση όπου εγώ είμαι η συγγήτρια στις 11 ε, θα παρουσιαστεί μια πολύ σημαντική έρευνα όποιοι δεν πρέπει να φύγουν θα παρακαλούσαν να παραμείνουν. Σας λέω λοιπόν εντάχει για την ε, δική μου παρουσίαση μιλάμε για την ισότητα των δύο φύλων ε, έναντι της φτώχειας. Όπως γνωρίζετε τα κείμενα πρέπει να είναι πολύ σύντομα και έχω θέσει έξι σημεία τα οποία μπορούμε να διευρύνουμε. Τα πιο σημαντικά ζητήματα σχετίζονται με μια βασική ε, ατζέντα του 2030 για να δούμε πώς τα παιδιά θα πρέπει να ορίσουν και να συμμετάσχουν σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και την φτώχεια στα, σε επίπεδο μικρών παιδιών. Έχουμε πολύ ε, ανησυχητικά στοιχεία γιατί ένα παιδί στα τέσσερα ε, διέπεται από φτώχεια. και υπάρχει και το θέμα στις υπηρεσίες για την υπιακή ε, ηλικία για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει σωστή, σωστός προσανατολισμός ως προς την επαγγελματική κατάρτιση, αν και ξέρουμε ότι πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση, σωστή πρόσβαση στην εκπαίδευση και αυτό που έχει σημασία είναι να ενισχύσουμε και τα δύο φύλλα έτσι ώστε να μπορούμε να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά την εκπαίδευση των μικρών παιδιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι έχει μεγαλύτερη σημασία ο τίτλος σπουδών των, της μητέρας παρά του πατέρα. Και πολλές φορές ε, η κατάρτιση της μητέρας στον τρίτο κόσμο έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τη διατροφική ασφάλεια. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις ε, μονογονεϊκές οικογένειες, τις ε, οικογένειες των προσφύγων, την ψυχική και σωματική υγεία και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε έτσι ώστε να μην υπάρχει εγκατάλειψη του σχολείου. Ένα θέμα που με απασχόλησε είναι να υπάρχουν ποιοτικά πρότυπα και προδιαγραφές για την ε, προσφορά εκπαίδευσης, ε, ιδιαίτερα ως προς τους μετανάστες και να εγγυηθούμε την εκπαίδευση και στους καταβλισμούς προσφύγων. Δυστυχώς 400.000 παιδιά πρόσφυγες στην Τουρκία δεν ε, καταρτίζονται, δεν ε, έχουν εκπαίδευση. Αυτό το είπαμε και στη Μογκερίνη, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα και εμείς την επόμενη Ολομέλεια. Και ξέρουμε ότι δυστυχώς τα κορίτσια υφίστανται και, και περαιτέρω διακρίσεις. Ε, τα αγόρια είναι αυτά που εγκαταλείπουν νωρίτερα το σχολείο, μαθαίνουμε. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφοροποίησεις ε, ανάλογα με τις επιλογές και ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο κόσμο της ε, πληροφορίας τα κορίτσια έχουν άλλες ε, δυνατότητες. θα μπορέσουν να υποβληθούν ε, τροπολογίες μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και στη ΦΑΜ στις 18 Απριλίου θα συζητηθεί το θέμα. Αν υπάρχουν παρεμβάσεις, έχουμε λίγο χρόνο, 6 λεπτά. Υπάρχουν μόνο δύο παρεμβάσεις, ε, Μωρέν Σαρτιέ και, Μορέν και Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξαίρετη η παρουσίαση του θέματος αυτού που ξέρω πόσο πολύ σας ενδιαφέρει εσάς και πάνω στο οποίο δουλεύουμε εδώ και χρόνια. Θέλω να μιλήσω για τρία σημεία σήμερα στην πρώτη συζήτηση. Το πρώτο έχει να κάνει με τον προσανατολισμό. Νομίζω ότι στην έκθεσή μας πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή βούληση προκειμένου ο επαγγελματικό ε, προσανατολισμός να σπάσει τα στερεότυπα ποια είναι η δουλειά για τα κορίτσια και ποια για τα αγόρια ή ποιε σπουδέ είναι για τα κορίτσια και ποιε σπουδέ είναι για τα αγόρια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Έχουμε κάνει πράγματα τα οποία έχουν δουλέψει καλά. Κάποια διαφήμιση που λέγαμε ότι α, είναι τεχνικές σπουδές ε, κάνουν για αυτήν. Ή ακόμα και στον οικοδομικό τομέα, που συνήθως πηγαίνουν τα γόρια, ενώ και τα κορίτσια μπορούν κάλλιστα να δουλέψουν εκεί, ακριβώς γιατί τα επαγγέλματα έχουν αλλάξει. Δεύτερον, Πιστεύω ότι η έκθεσή μας πρέπει να είναι σαφής και ως προς το Στην παράγραφο 6, στο σημείο 6, αναφέρεστε στις... Ε, ότι λέτε μάλλον ότι τα αγόρια πολύ πιο συχνά δεν έχουν δίπλωμα, ενώ τα κορίτσια ναι. Δηλαδή, κάνοντα σπουδέ δεν καταλήγουν σε κάποιο δίπλωμα τα αγόρια. Με αυτό και εδώ διαφωνώ μαζί σας, πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Ένα αγόρι που βαριέται στο σχολείο, συμπεριφέρεται αλλιώ. Και πολύ εύκολα του δείχνουν την πόρτα. Ενώ το κορίτσι αν βαριέται, αναδιπλώνεται, δεν εκδηλώνεται και παραμένει στην τάξη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας οι δάσκαλοι δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν έχουν να κάνουν με ένα γόρι που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο από ότι με ένα κορίτσι. Γι' αυτό και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το τρίτο σημείο τώρα έχει να κάνει με κάτι που το αναφέρεται μεν, αλλά ίσως όχι αρκετά. Τις επιπτώσεις που έχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες πάνω στα παιδιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα αυτό. Οι μονογονοϊκές οικογένειες, όπως και άλλες, δεν αποκλείεται, καταλαβαίνετε, ο γονιός αυτός να αρρωστήσει. Και καρκίνο ή το οτιδήποτε που απαιτούνται μεγάλες θεραπείες. Τότε τι γίνεται, ο προστάτης γίνεται το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης και σπουδών. Και αντίθετα, έχει περισσότερες πιθανότητες να καταλήξει στη φτώχεια από ό,τι άλλοι. Γι' αυτό πρέπει να προβλέψουμε πώς θα διορθώνουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέροντα όσα αναφέρατε. Θα τα λάβω υπόψη. Η κυρία Evans και μετά Διάκονο, ο κύριος Διάκων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την έκθεση αυτή. Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία που θίξατε. Αγαπητοί συνάδελφε, η φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό φυσικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τι γυναίκες. Είναι μια τάση που επιμένει μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να γίνει αναφορά στην παράγραφο 4 για τις ε, μονογονεϊκές οικογένειες. Το 85% των μονογονεϊκών οικογενειών ε, ε, είναι με γυναίκες ε, στην κεφαλή της οικογένειας, οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση και χρειάζονται λοιπόν ε, επιγόντως την ε, βοήθειά μας. Τώρα, σίγουρα τα κορίτσια έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις, όμως αυτό δεν διαφαίνεται στον εργασιακό τομέα, στην αγορά εργασίας. Και πιστεύω πως πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτό. Επίσης, πιστεύω πως τόσο η εκπαίδευση όσο και ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και η εκμάθηση γλωσσών, διότι η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ε, και αυτή συνδεδεμένη με την ε, γνώση ξενών γλωσσών. Και πρέπει να προσέξουμε να ε, μην αποκλείονται οι νέοι με αυτόν τον φαύλο κύκλο, όπως είπατε, και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες. Επίσης πιστεύω πως πρέπει να γίνει μια αναφορά στο, στα όσα έχουν ήδη γίνει, στην δουλειά που έχει γίνει από διάφορους οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει ένα, μια οργανώση που λέγεται Fair Play, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιείται κυρίω στην καταπολέμηση των ε, στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που έχουν ε, οι άνθρωποι και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών. Πιστεύω λοιπόν πως πράγματι η εκπαίδευση πρέπει να λάβει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην έκθεση αυτή και μπορούμε να την βελτιώσουμε την έκθεση κάπως. Γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλω τις δικές μου προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ε, Διάκονου και μετά θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή αν έχει κάτι να πει. Θεωρητικά και μόνο θεωρώ ότι ε, οι βοηθοί μας θα πρέπει να μπορούν να μας βοηθήσουν καλύτερα και εάν οι βοηθοί μας είναι περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες, ε, όπως και οι διερμηνείς, σημαίνει ότι η κυρία Σίλβια έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι αλήθεια, δεν, είναι, δεν το παγιαστείο. Τώρα για να σοβαρευτούμε και λιγάκι, θεωρώ ότι η φτώχεια είναι μεγάλο δράμα. Όταν μιλάμε για παιδιά ιδιαίτερα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξαλειφθεί η φτώχεια στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή θέλει κάτι να πει. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σημειώσαμε κάποιες ε, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που υποβάλλεται και στο κείμενο αλλά και όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στις ε, γραπτές προτάσεις του κεφαλαίου για την εκπαίδευση και την ε, μέρημνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Επίσης επηρεάζει πολύ την συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας διότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ε, καμιά φορά ε, ένα σημαντικό εμπόδιο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γνωσιακή ανάπτυξη των ε, παιδιών και για να διασφαλίσει την επιτυχημένη ε, ένταξή του στην αγορά εργασίας ε, στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένως προσπαθεί να στηρίξει όσο μπορεί τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τα παιδιά. Βέβαια, σημειώνουμε και το γεγονός ότι εσείς αναφέρεστε σε αυτό στο κείμενο και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι μια πρόκληση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, την παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα προσπαθήσουμε επίσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να ε, δημοσιεύσουμε συστάσεις. Βασίζομαι στη συνεργασία σας και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ε, συνεισέφεραν έμπρακτα επί του θέματος. Θα συνεργαστούμε και θα ήθελα να πω ότι στις 18 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τις 3. Περνάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, καλεσμένους. Μόλις ε, έφτασαν εδώ, ευχαριστώ τους ερευνητές Έχουμε μια αντιπροσωπεία επισκεπτών από τη Γαλλία, διευθυντών και επιθεωρητών σχολείων από τη Μπουργκόνια ε, υπό τον Εντουαρ Μαρτέν του Σεντίκ ε, το θέμα είναι άκρος ε, ενδιαφέρον που θα παρουσιαστεί. Η Επιτροπή Πολιτισμού συνεισέφερε στην κατάρτιση αυτής της έρευνας και νομίζω ότι το θέμα αυτό ανέκυψε και από τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Eh, eh, γνωρίζετε ότι στόχος είναι να ε, υπάρχει κριτική ανάλυση του θέματος ε, της ε, διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι μια πολύ καλή βάση για να δούμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία αυτής της μελέτης και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά για μια βαθύτερη γνώση των συνιστοσών του ζητήματος. θα θέλαμε να ε, ανακύψουν και συστάσεις και απότερες στρατηγικές. Η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί από την κυρία Φιώνα Χάντερ από το Center for Higher Education Internationalization του Università Κατόλικα του Μιλάνου και την κυρία Εύα Γκρον Πολάκ της ε, IAU του Παρισιού, από το Παρίσι. Θα βλέπετε και τις διαφάνειες και θα σας δώσω τις κατάλληλες πληροφορίες στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που είναι παρόντες. Το έγγραφο αυτό θα κοινοποιηθεί σε όλους και θα, γίνουν, θα υπάρξουν συνεχείς επαφές επί του θέματος. Δεν ξέρω ποια θα μιλήσει πρώτα. Λοιπόν, η κυρία Χάντερ. Καλημέρα σε όλους. Θα σας κάνω εγώ την παρουσίαση σήμερα το πρωί και η συνάδελφός μου η Εύα θα σχολιάσει κάποιες από τις διαφάνειες. Και θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη, διότι πρέπει να φύγω στις 12 και 20. Πρέπει να πετάξω προς την Μαλαισία και αυτή την πτήση την είχα προγραμματίσει πριν ε, προσκληθώ να έρθω εδώ. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρω να προλάβω, να είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Όμως η Φιώνα είναι η ε, κύρια παρουσιάστρια της μελέτης και θα είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω, εάν δεν έχετε διαβάσει τη μελέτη, ότι το βασικό ερώτημα που κληθήκαμε να απαντήσουμε είναι το εξής. Ποιες είναι η, ε, ποια είναι η ουσία της εσωτερικοποίησης και πού πρέπει να στοχεύουμε. Αυτή η παρουσίαση θα προσπαθήσει να συνοψίσει με λίγες διαφάνειες ε, το ερώτημα αυτό σε δύο τμήματα. Καταρχάς θα κοιτάξουμε ε, τι ξέρουμε μέχρι τώρα και ποια νομοθεσία υπάρχει και ε, θα εστιάσουμε κυρίως στην Ευρώπη σε αυτό και στη μελέτη μάλιστα. Εστιάσαμε και σε κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στο δεύτερο δε μέρος της μελέτης θα ρωτήσουμε τι θα έπρεπε να ε, θέλουμε, σε τι θα έπρεπε να στοχεύουμε, ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική μας κατεύθυνση. Θα γίνουν μερικές προτάσεις που επικεντρώνονται κυρίως στο ότι η κατεύθυνση στην οποία οδεύουμε δεν είναι αυτή που θεωρούμε ως ε, καταλληλότερη για την Ευρώπη. Ένα από τα σημαντικότερα ε, πορίσματα που προέκυψαν από τη μελέτη είναι ότι η εσωτερικοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ νέο. Είναι ένα νέο φαινόμενο και μια νέα λέξη, νεολογισμός έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα αν σκεφτείτε, πολλοί από εμάς δεν είχαμε ακούσει αυτόν τον όρο μέχρι τώρα και δυσκολευόμαστε μέχρι και να τον προφέρουμε. Αφορά λοιπόν χώρες ε, και θεσμικά όργανα. Δυστυχώς υπάρχει μια ευρύτατη έννοια της εσωτερικοποίησης και δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να μπορούμε ενιαία να ακολουθήσουμε. Η εσωτερικοποίηση είναι ένας όρος που αλλάζει συνεχόμενα και επηρεάζεται από ένα ευρύτατο φάσμα ε, απόψεων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών. Και τονίζω την οικονομική διάσταση διότι είναι η επικρατούσα τάση στην εσωτερικοποίηση. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μία τάση για την ιδιωτικοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης και επομένως η εσωτερικοποίηση ταυτίζεται λέω, και περισσότερο με το κέρδος αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ευρώπη, αν και υπάρχει ίσως μια εξαίρεση για ορισμένες χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, είναι ότι υπάρχει μια μετατόπιση στην εσωτερικοποίηση, ε, όπως στην, ε, μάλλον διάσταση του ανταγωνισμού. Υπάρχει μια μεταστροφή προς τον ανταγωνισμό και η μελέτη αυτή κοιτάζει το ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα η εσωτερικοποίηση και προσπαθεί να εξετάσει την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής. Ε, εμείς ως ε, Διεθνής Ένωση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προσπαθήσαμε να κοιτάξουμε τις ε, παγκόσμιες τάσεις και να εξετάσουμε τις διάφορες μελέτες και τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την κάθε χώρα ξεχωριστά. Και σταθήκαμε επίσης και στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορες χώρες, πολλές εκτός Ευρώπης που δεν έχουν το πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής αγοράς, μιας ευρωπαϊκής αγοράς που είναι πολύ πιο συνεργατική σε σχέση με την Ασία ή με τη Βόρεια Αμερική. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ εντονότερο και αυτό είναι και γνώμονας της ε, εσωτερικοποίησης της διαδικασίας αυτής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε. Μία άλλη επικρατούσα τάση είναι ότι γίνεται όλο και σημαντικότερο στρατηγικά. Ε, και σε κρατικό και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο παρατηρείται μία τάση, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής, προς μία πιο ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση στην εσωτερικοποίηση. Βλέπουμε πως ε, διεθνώς αναπτύσσονται στρατηγικές εσωτερικοποίησεις και αυτό φαίνεται εντονότερα σε χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα έντονες εθνικές βλέψεις και φιλοδοξίες. Η εσωτερικοποίηση λοιπόν συνδέεται άμεσα με το, την εθνική ατζέντα κάποιας ε, χώρας και όσο υψηλότερα είναι στις προτεραιότητες της χώρας αυτής ε, τα ε, εθνικά συμφέροντα, τόσο και η εσωτερικοποίηση θα είναι πιο συνδεδεμένη με αυτά. Υπάρχουν εσωτερικές στρατηγικές για την εσωτερικοποίηση λοιπόν και ε, αναπτύσσονται όλο και περισσότερα μοντέλα και στρατηγικές εσωτερικοποίησης. Αυτό που παρατηρούμε σε όλα αυτά τα μοντέλα είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα προγράμματα, μεγαλύτερη κινητικότητα, γενικότερα περισσότερη δράση. Βλέπουμε Δηλαδή ότι η στρατηγική βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές ε, χώρες ε, πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία δυσκολεύονται διότι κυρίως ε, τους λείπουν τα σωστά ε, στοιχεία για να λάβουν αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι κυρίως σε εθνικό επίπεδο και όχι διασυνοριακά. Επίσης βλέπουμε την μεγαλύτερη περιφερειακή διάσταση της εσωτερικοποίησης. Οι χώρες κοιτού, κοιτάζουν προς τις γειτονικές τους χώρες, προς τις περιφέρειες και εστιάζονται ε, σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μοντέλο που αναδύεται είναι πιο περιφερειακό και κυρίως ευρωπαϊκό από ό,τι παρατηρούμε. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε. Πιστεύω πως αν τα κοιτάξει κανείς είναι σαφές ότι ε, τα στατιστικά στοιχεία αφορούν περισσότερο την κινητικότητα γιατί είναι εύκολα μετρήσιμη. Και μπορούμε να δούμε λοιπόν ε, πιο ε, προσεκτικά την κινητικότητα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εσωτερικοποίησης. Υπάρχουν όμως και άλλες διαστάσεις ε, της ε, διαδικασίας αυτής και κάποια άλλα πιο δύσκολα μετρήσιμα ε, νούμερα, τα οποία επηρεάζουν όμως εξίσου τόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και τους σπουδαστές. Γι' αυτό λοιπόν δεν αρκεί να κοιτάζουμε μόνο τους σπουδαστές. Έπειτα όσον αφορά την ε, περιφερειακή διάσταση πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα μάλιστα αν κοιτάξουμε τι γίνεται και στις άλλες υπήρους, στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Ασία. Εκείνες οι ήπειροι θεωρούν το ευρωπαϊκό μοντέλο ε, ως ε, παράδειγμα προς μίμηση, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κινητικότητας και της αναγνώρισης των πρακτικών. Δεν μιλάω μόνο για το πρόγραμμα Εράσμους, αλλά και για τις ευρύτερες δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα για να προωθήσει την εσωτερήκευση. Όλα άρχισαν λοιπόν από το Εράσμους. Πιστεύω πως ε, αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μοντέλο μαζί με, την, ε, με τις ε, μεταρρυθμίσεις της διαδικασίας της Μπολόνια άλλαξε τα δεδομένα και έγινε η κινητήριος δύναμη της εσωτερικοποίησης. Όπως ε, ακούστηκε, επηρέασε πάρα πολύ σημαντικά και άλλες περιοχές του κόσμου και γι' αυτό παρατηρείται αυτή η τάση της συνεκτίμησης ε, της εσωτερικοποίησης, εσωτερικοποίησης στην ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης, ε, πολλά λέγονται για την εσωτερικοποίηση, όμως διεθνοποίηση. Βλέπουμε πως ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί στην Ευρώπη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα στη μελέτη μας σε παγκόσμιο επίπεδο για τις προκλήσεις είναι το εξής, ότι ακόμα και στην Ευρώπη που είναι η πιο προηγμένη ήπειρος σε αυτό το θέμα, υπάρχει πρόβλημα στην αναγνώριση σπουδαστικών ε, μονάδων και περίοδους φίτησης. Είναι ένας κίνδυνος που προστίθεται στους άλλους κινδύνους. Και βλέπουμε ότι η διεθνοποίηση είναι δηλαδή διαθέσιμη μόνο σε όσους μπορούν να την αντέξουν οικονομικά. Η πρόσβαση λοιπόν Και η κινητικότητα είναι κάτι που στην εθνοποίηση είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τα θεσμικά όργανα. Και όπως είπε και η Φιώνα, έχει επηρεάσει αυτό διαφορετικά την κάθε περιοχή στην Ευρώπη. Βλέπουμε το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βλέπουμε δηλαδή ότι οι σπουδαστές, φοιτητές, απόφοιτοι εγκαταλείπουν τις ε, χώρες τους και πηγαίνουν αλλού. Και αυτό είναι μια πρόκληση όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για άλλες υπήρους όπως την Αφρική για παράδειγμα. Βλέποντας λοιπόν πώς αυτό το δυναμικό επηρεάζει τα δεδομένα στην Ευρώπη, υπάρχουν διάφορα μοντέλα που αναδύονται, τα οποία τείνουν να επικεντρώνονται σε αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς. Καταρχάς, υπάρχει η βραχυπρόθεσμη, η μακροπρόθεσμη διάσταση του κέρδους, δηλαδή οι σπουδαστές προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, κερδοφόρες ε, σχέσεις για το μέλλον τους, υπάρχουν ε, διάφορες επιχείρησεις που δραστηριοποιούνται έτσι ώστε να ε, βοηθήσουν στην εύρεση εργασία, στην ορατότητα κάποιου εργαζόμενου και επίσης όσον αφορά την ορατότητα η ευρωπαϊκή αγορά έχει δώσει πάρα πολύ έμφαση στην κινητικότητα και τη θεωρεί ένα πολύ βασικό ε, στοιχείο της εθνοποίησης. Τώρα, πώς ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Πιστεύουμε πως χρειάζεται μία πολύ πιο συνολική προσέγγιση και πολύ πιο συνεκτική, ίσως αυτή είναι η καλύτερη λέξη, σε θεσμικό επίπεδο πρέπει η διεθνοποίηση να είναι πάρα πολύ σημαντική και προσαρμοσμένη στις ε, ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει μία ε, λύση για όλους. Η κινητικότητα σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, όμως αν πραγματικά θέλουμε να ε, δώσουμε πρόσβαση στη διεθνοποίηση, πρέπει να εστιάσουμε στη διδακταία ύλη. Πρέπει να δούμε τι μοντέλο θέλουμε να δημιουργήσουμε, τι είδους ε, παγκόσμιο πολίτη θέλουμε να έχουμε και μετά να δούμε πώς εκείνος μπορεί να δραστηριοποιηθεί παγκόσμια, πώς μπορεί να βρει δουλειά ε, παντού στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο πρόγραμμα, στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, προγραμματισμός και διδακτάιλη. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να υπογράψουμε για άλλη μια φορά είναι το πιο ευρύ επίπεδο από το ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για το 20%. Που σημαίνει ότι το 80% των ε, υπόλοιπων ε, φοιτητών δεν θα πάει πουθενά αλλού πέρα από εκεί που σπουδάζει. Και μόνο το 3% φοιτών έχει τη δυνατότητα αυτή. Αν λοιπόν κοιτάξουμε το πρόγραμμα, το σχολικό, αν δούμε τι μαθαίνουν τι έρευνες κάνουν στην ανώτατη εκπαίδευση οι φοιτητές, η διεθνής διάσταση θα αγγίξει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει η σύνδεση αυτή της διεθνούς ε, διάστασης με τις σπουδές γιατί μόνο τότε εξυπηρετούν οι στόχοι της ανώτατης ε, εκπαίδευσης. Δεν είναι αυτός σκοπός, πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους της εκπαίδευσης. Και όντως καταφέρνει και αντιμετωπίζει κάποιες από τις προκλήσεις των σπουδών που είναι έτσι καλλιώς διεθνείς, εξορισμού. Είναι κλειστό το μικρόφωνο της ομιλήτριας, δεν την ακούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό και πάμε πιο γρήγορα τώρα στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης. Στη μελέτη αυτή πολλά θα σας ε, εξηγήσουν πώς εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και ένα τμήμα της μελέτης είναι ότι κοιτάξαμε ποιος είναι ο πιο αποδεκτός ορισμός της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε όμως τον ορισμό και θα ήταν ε, ένα καλό σημείο κίνηση. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, αλλά α πούμε ότι ένα που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι εκείνο του James Knights, που λέει ότι η διαδικασία ολοκλήρωση μια διεθνού διαπολιτιστική και σφαιρική διάσταση στου σκοπού ε, και τη λειτουργία και τα αποτελέσματα τη ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Είναι ορισμό που χρησιμοποιείται τα τελευταία 10-15 χρόνια ανοίγει ευκαιρίες για να μπορέσει ο καθένας να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης. Εμείς επικεντρωνόμαστε πάντως σε αυτόν τον ορισμό και έχουμε προσθέσει σε αυτόν την ε, ε, με σκοπό τέτοια διαδικασία ολοκλήρωσης μιας ε, διεθνούς διαπολιτισμικής και σφαιρικής διάστασης. Και εξηγούμε και γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για να ενισχύσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας για όλους τους μαθητές και το προσωπικό και για να συνεισφέρουμε έτσι ουσιαστικά στην κοινωνία. Λέει ότι είναι μία διαδικασία που γίνεται με σκοπό. Πρέπει δηλαδή να έχει νόημα για τη δικιά σας την αποστολή. Να λάβετε υπόψη σας το τι θέλετε σημαίνει ότι θα το επιλέξετε, ότι θα το αποφασίσετε και θα δράσετε. Δεν πρόκειται μόνο για λόγια. Πρόκειται και για πράξεις. Εμείς τη διεθνή διάσταση της ε, ανώτατης εκπαίδευσης την βλέπουμε σε κάτι που πρέπει να βοηθήσει να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι σε αυτή. Βασική διάσταση είναι ότι πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ε, σχολικού, μάλλον ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους. Πρέπει όλος ο ακαδημαϊκός ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει διεθνή διάσταση εκπαίδευση. Την διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης λοιπόν δεν πρέπει να τη δούμε σαν έναν αυτό σκοπό, αλλά για να βελτιωθεί η ποιότητα και για να συνεισφέρει στην κοινωνία. Και ενώ το οικονομικό στοιχείο θα παραμένει πάντα, αυτό που εμεί λέμε είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στο οικονομικό κέρδος μέσω της διεθνούς αυτής διάστασης της εκπαίδευσης. Και θα αφήσω τη συνάδελφο να ολοκληρώσει. Ναι, ο ορισμός αυτός λοιπόν της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης έχει πετύχει συνένεση. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Δεν είναι βέβαια κάτι ουδέτερο. Υπάρχουν ε, λόγοι και πέρα από τον ακαδημαϊκό. Ο νέος λοιπόν ορισμός αναφέρεται στον σφαιρικό στόχο που δεν είναι καταρχήν οικονομικός, είναι καταρχήν ακαδημαϊκός και επιστημονικός. Γι' αυτό και είναι πιο χρήσιμος ο ορισμός, πιο κατάλληλος, που μπορεί βέβαια να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί ανάλογα με τις επιπτώσεις που έχει η διεθνοποίηση εκπαίδευση στην ποιότητα και στην αντιμετώπιση τοπικών και σφαιρικών ζητημάτων. Και ένα τελευταίο μου σχόλιο. Η Ευρώπη έχει μια τεράστια ευκαιρία αλλά και τεράστια ευθύνη, ακριβώς γιατί όλοι την κοιτούν ως μοντέλο είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να αντικατοπτρίζουν αυτές τις σημαντικές αξίες της ανώτατης εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθών. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακριβώς η Ευρώπη, εκτός από το ότι αποτελεί αντικείμενο για τους άλλους, η ίδια πρέπει να κοιτάει προς τα έξω. Είναι δηλαδή δύο διαδρομών η διαδικασία αυτή, δύο κατευθύνσεων, και η Ευρώπη κοιτάει προς τα έξω για να παραδειγματιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλούσια έρευνα γιατί μας ε, αποστέλει ένα βασικό μήνυμα, δηλαδή να ξανασκεφτούμε το θέμα της διεθνοποίησης της ε, διαδικασίας της εκπαίδευσης. Σε αυτή τη φάση εκκίνησης προγραμμάτων ε, διεθνοποίησης και μετά την διαδικασία της Μπολόνια, θα πρέπει μέσω της δικής σας εργασίας, όπου συμμετείχαν 17 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, αυτό που θα έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε τη διπλή αυτή πρόκληση. Καταρχήν πώς να ε, θεσμοθετήσουμε τη συμμετοχή σε προγράμματα. Το Erasmus είναι ένα από αυτά. Και το άλλο θέμα είναι το άνοιγμα, η έναρξη ενός διαλόγου με τα πανεπιστήμια, γιατί μας ενδιαφέρει να διεθνοποιήσουμε την εμπειρία αυτή, όχι μόνο έξωθεν, με βάση έξωθεν δεδομένα, να ενισχύσουμε το, το, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις οικονομικές ευκαιρίες, μία ευρύτερη θεώρηση των θεσμών και μία επένδυση στους ανθρώπους μέσα στα πλαίσια μίας ισότητας πέρα από την ποιότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για μία ε, σελίδα, καινούργια σελίδα που ανοίγει πέρα από τα ιωθώτα και του τι αναφέρεται γενικότερα σε αυτό το τομέα, θέλαμε να ε, διασφαλίσουμε το διπλασιασμό των πόρων του Erasmus Plus για τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά δεν ε, δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αυτό να το ξέρουμε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες αυτές ε, προοπτικές, θα ήθελα πριν να σας δώσω το λόγο ότι υπάρχει και άλλη μια ομάδα επισκεπτών, 15 επισκέπτες από την ε, Ένωση Εκπαιδευτικών ε, από τη Σουηδία, ε, είναι από την ομάδα των Πρασίνων και τους έχει προσκαλέσει ο βουλευτός μας ο κύριος Άντερσον που ήσασταν εκεί στο, στο βάθος της αίθουσας. Θα δώσω το λόγο σε όσους τον ζήτησε. Σο, Σοϊντρόβα, Βέντα, Μόργανο, εντάξει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομιλήτριές μας για την παρουσίαση αυτή. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να την μελετήσω σε βάθος. Φοβάμαι πάντως ότι για να τη χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς μας σκοπούς, για να συζητήσουμε το Erasmus ΣΥΝ, για παράδειγμα, να το χρησιμοποιήσουμε για να συντονίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που χρειαζόμαστε είναι τον έλεγχο του τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αυτή η επιλεκτική μελέτη φυσικά είναι εφικτή, αλλά για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε υπεύθυνα την κατάσταση, χρειαζόμαστε μια πιο γενική μελέτη. Και θέλω να σας ρωτήσω τη γνώμη σας από αυτού. Τώρα και οι δυο σα αναφερθήκατε στον κίνδυνο διαρροής εγκεφάλων. Πράγματι, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει κυρίως τις νέες χώρες μέλη, γιατί οι φοιτητέ ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να πάνε σε ένα γνωστό μεγάλο πανεπιστήμιο. Είναι όμως κάτι που βελτιώνεται, πιστεύω. Και θέλω να επιβεβαιώσω εδώ ότι τα διορθωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποίησαμε για να φτιάξουμε επιστημονικά κέντρα σε περιφερειακά πανεπιστήμια στην Τσεχία, παρόλο που έχουν βέβαια κάποια προβλήματα να κρατήσουν τον κόσμο, παρόλο, παρόλο αυτά τα κέντρα αυτά ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία, γιατί γίνονται κέντρα αριστείας στον τομέα τους και ως τέτοια μπορούν να καλύψουν τους στόχους της διεθνοποίησης που αλλιώς δεν μπορούν να το κάνουν. Τα διευθυντικά ταμεία μπορούν να χρησιμεύσουν λοιπόν. Αλλά ξέρω ότι τα κέντρα αυτά και σε άλλες χώρες και στην Ουκρανία φοβούνται αυτή τη διαρροή εγκεφάλων και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Εσείς θα μπορούσατε να σχολιάσετε Πώς να αντιμετωπίσουμε τη διαρροή εγκεφάλων διατηρώντας τη διεθνοποίηση. Πέρα από τα οικονομικά μέσα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, πρέπει να έχουμε και υψηλή ποιότητα σε εκπαιδευτέ στην ανώτατη εκπαίδευση, να πληρώνονται καλά και έτσι να προσελκύουν ε, φοιτητέ. Είναι σίγουρα οικονομικό το ζήτημα πρέπει να διασφαλιστούν τα οικονομικά των πανεπιστημίων, κυρίω στην, στην Ήπετρο, εκεί που έχουμε πανεπιστήμια που δεν είναι τόσο γνωστά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βέντα. Η συνάδελφος είπε πολλά από αυτά που σκόπευα και εγώ να πω. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ξέρω ότι βιαζόμαστε, οπότε μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μιλάτε για τη διαρροή εγκεφάλων. Έχετε νούμερα που μπορείτε να μας δώσετε για να καταλάβουμε περίπου πόσοι φεύγουν και τι, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε τους νέους στην Ευρώπη. Έπειτα έχουμε δει ότι το υλικό είναι ευρύ. Έχουμε το Εράσμος, από εκεί ξεκίνησαν εξάλλου όλα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε περισσότερο και να δούμε και τους ορισμούς. Πάντως όσα μας είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα κυρίως για το επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ας δούμε τα νέα κράτη-μέλη, τη δικιά μου τη χώρα, για παράδειγμα εκεί, αυτό που είναι βασικό είναι η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, ανώτατης εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένα νούμερα και εδώ, γιατί είναι πρόκληση για πολλούς και τι γίνεται, όταν τελειώσει κανείς την εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανώτατη εκπαίδευση δηλαδή, και έχει το δίπλωμά του, μετά τι γίνεται. Για να μπορούμε να έχουμε και στο περιφερειακό επίπεδο κάτι και όχι μόνο στο διεθνές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μόργκανο, Μόργανο, ε, λέγοντας ότι αυτή η εξαιρετική έρευνα βρήθη στοιχείων και θα σας ζητήσουμε και άλλες διευκρινήσεις αν ανακύψει λόγος γιατί πρόκειται για έναν μεγάλο πλούτο. Ε, το iVersity ε, μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή η θεματική αυτή που προβάλλεται και νομίζω ότι μας εμπλουτίζει ιδιαίτερα γιατί αυτά τα οποία μας απασχολούν ήδη ενσωματώνουν στο κείμενο. Λουίτζι, ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ καταρχήν για την εισήγησή σας. Ακόμα δεν έχουμε ε, αναγνώσει το κείμενο, αλλά έριξα μια ματιά και βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε μία συγκριτική μελέτη ή συγκριτική ανάγνωση με βάση τα πράγματα πώς, ε, ως προς το πώς έχουν σήμερα. Έχουμε λοιπόν τις ε, συνολικές τάσεις αλλά και μία εσωτερική ανάγνωση για να δούμε πώς έχει το θέμα στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιδράσουμε επί της ουσίας. Νομίζω ότι υποστηρίζεται κάτι το απόλυτα σαφές. Θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε αυτή τη διεθνοποίηση. Δεν είναι θέμα μόνο κινητικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μεγάλα βήματα ε, είναι σαν να μιλάμε για ένα στόχο που χρειάζεται ορισμένους επιμέρους στόχους ή στοχοθετήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε και με το θέμα της απασχολησιμότητας, αλλά δεν μας ορίζει το μέλλον μόνο ένα οικονομικό ή πολλά οικονομικά στοιχεία γιατί θα μπορούσαμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τις δυσκολίες και να επιτρέψουμε την συμμετοχή στην ε, αγορά εργασίας. Τώρα, ως προς την ε, ποιότητα, αυτό είναι ένα αναπόδραστο στοιχείο. Και εδώ μιλάμε για μία γενικότερη σκέψη που αφορά τον ακαδημαϊκό κόσμο. Γιατί γι' αυτόν ε, μιλήσατε αρχικά. Και αυτό σημαίνει κατά τη δική μου άποψη και θέλω διευκρινήσεις επ' αυτού ότι θα πρέπει να υπερβούμε την προσέγγιση των μεμονωμένων κρατών κάτι το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με την αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δέχομαι αυτή την ε, πολιτισμική πρόκληση και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί μόνο το 3% αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να καρποθεί μια τέτοια ευκαιρία. Αυτό είναι το αντικειμενικό στοιχείο που διαθέτουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτές τις ε, δυνατότητες, κάτι το οποίο ε, είναι ουσιώδες. Τώρα πέρα από τη διαδικασία της Μπολόνια που έγινε στο Ερεβάν. Α, εντάξει, εσείς μπορείτε να φύγετε. Ε, εσείς μπορείτε να πάτε στη Μαλαισία ανεξάρτητα από τη δική μου παρέμβαση. Μπορείτε να αποχωρήσετε. Το θέμα είναι στα προγράμματα σπουδών να δούμε τι μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή παρά την ε, ε, νομική υπόσταση των τίτλων σπουδών. Είναι κάτι το οποίο ε, πλαισιώνει αυτή την έρευνα και η επιστημονική έρευνα είναι πιο ευρεία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας σας ε, δίνω το λόγο για να μπορέσετε να φύγετε για τη ε, Μαλαισία και θα ήθελα να τονίσω ότι συμμετείχαν 17 χώρες, 10 ευρωπαϊκές και 7 μη ευρωπαϊκές, μεταξύ των οποίων και η Μαλαισία. Answer you fully, but I... Ευχαριστώ πολύ. Ε, ίσως να μην καταφέρω εγώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά η Φιώνα θα το κάνει σίγουρα. Ε, διαρροή εγκεφάλων. Σίγουρα υπάρχουν ε, πάρα πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλά θεσμικά που που τραβάνε τους εγκεφάλους, τους νέους εγκεφάλους, νέους επιστήμονες. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε περισσότερο είναι πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, γιατί ξέρω ας πούμε πως στην Τσεχία υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Πράγας και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα που ε, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση έτσι ώστε αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να διατηρήσουν ε, την ε, ελκυστικότητά τους στους φοιτητές. Ε, και χρειάζεται επίσης να φροντίσουμε για την πληροφόρηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σωστή ιεράρχηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και να αποτραπεί τα πιο γνωστά να βλάψουν την φήμη των λιγότερων γνωστών, των μικρότερων. Αυτό που πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι χρειάζεται να συνομιλήσουμε περισσότερο και καλύτερα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρά με την πολιτική. Βέβαια η μελέτη αυτή αφορά κυρίως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτό φαίνεται και στην έκθεσή μας. Αυτό όμως που βλέπουμε στο χώρο της πολιτικής είναι ότι οι εθνικές πολιτικές ε, διαφοροποιούνται. Ε, υπάρχει η εθνική στρατηγική που χαρακτηρίζονται ίσως από περισσότερη κινητικότητα, από περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να τραβήξουν φοιτητέ από, γεωγραφ, από την γεωγραφία, από το που βρίσκεται το κάθε ίδρυμα και από την άλλη από τον πραγματικό σκοπό ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, δηλαδή να υπηρετήσει τη μάθηση, τη γνώση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτός ο διαχωρισμός Πιστεύω πως η έκθεση υιοθετεί μία περισσότερο μεικτή προσέγγιση. Και λυπάμαι που πρέπει να φύγω, αλλά ε, θα τελειώσω εδώ. Και καλή πτήση να έχετε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η συναδελφός μου και στα σχόλια που κάνατε. Καταρχάς η προσέγγιση που προτείνουμε εμείς είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία. Και δίχως αμφιβολία, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στο πώς αντιμετωπίζουμε τη διεθνοποίηση, πρέπει να αλλάξουν πολλά, να αλλάξουν πολλά μακροπρόθεσμα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διεθνοποίηση, διότι αυτή ε, εκθέτει τις αδυναμίες των ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να κρατήσουμε ταυτόχρονα τα πάντα όπως ήταν και από την άλλη να προχωρήσουμε στη διεθνοποίηση. Πρέπει να ενσωματώσουμε τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποιότητα και η ικανότητα ε, και αποστολή αυτών των ε, ιδρυμάτων. Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα και να αφήσουμε τις θεωρίες κατά μέρους και όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή όποια κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει αυτές τις ε, προϋποθέσεις, αυτήν την ε, διαδικασία υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, πολλά εργαλεία, τρόποι, πρακτικοί τρόποι προσέγγισης. Υπάρχουν λοιπόν ε, τρόποι για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας τη διδακτέα ύλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφοροποιημένα μοντέλα κινητικότητας. Το εξάμεινο εξωτερικού, για παράδειγμα, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο ε, και βοηθάει πολύ μεν ατομικά, όμως είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί Ευρύτερα, επίσης, αν ε, καταφέρουμε να εισαγάγουμε στη διδακτέα ύλη κάποια στοιχεία διεθνοποίησης, η κινητικότητα είναι μεν ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί αυτή, δεν είναι όμως πανάκια και δεν μπορεί να συμπληρώσει τα κενά τα οποία δημιουργούνται από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, ε, να πούμε ότι αν υπάρχει ένα διεθνοποιημένο ε, σύστημα εκπαίδευσης, ε, μια διεθνοποιημένη διδακτέα ύλη θα επηρεαστεί με θετικό τρόπο και η κινητικότητα. Διότι όταν η κινητικότητα είναι ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος ε, που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και οι φοιτητές ε, την ε, μάθηση και την έβραση εργασίας αργότερα. Και πιστεύω πως η επιτυχία του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος έχει να κάνει με την πολυμορφία της. Η Ευρώπη έχει πάρα πολύ καλή φήμη εκπαιδευτικά σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την διεθνοποίηση λοιπόν έτσι ώστε να βοηθήσουμε και να γίνουμε το ε, παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης συνέργειες, όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους κλάδους. Και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας. Σας ευχαριστώ και για το ευρωπαϊκό σας όνειρο το οποίο συμμεριζόμαστε. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες στην οποία συμμετείχαμε και σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Θα ήθελα να τη διαβάσετε όλοι γιατί αποτελεί και ένα γνωστικό αντικείμενο ύψης της σημασίας. Ε, μιλήσατε για το θέμα της ολοκλήρησης, ε, αλλά το «Iversity» Ε, και το πώς τα πανεπιστήμια online μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν μια άλλη ποιότητα. Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση και φυσικά υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με την ε, διεθνή κινητικότητα, αλλά δεν ε, προβαίνουν σε μία σύγκληση για να ε, εντατικοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών, πέρα από την φυσική κινητικότητα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και είναι πολύ ενδιαφέρον διότι αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Δύο χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνέταξε μία ανακοίνωση για την ε, ανώτατη εκπαίδευση στον κόσμο που αποτελεί ένα κείμενο στρατηγικής και επειδή έχουμε τους ίδιους εμπειρογνώμονες τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με αυτά της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση ε, συντάχθηκε όταν ε, ξεκίνησε το πρόγραμμα ε, Erasmus Sin. Η κυρία Πόλακ είπε ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για διεθνοποίηση, αλλά θα πρέπει και να το προωθήσουμε έμπρακτα. Αυτό κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια με το Erasmus ΣΥΝ» γιατί πολλοί έχουν την ε, ε, εντύπωση ότι το Εράσμους ΣΥΝ ασχολείται με θέματα κινητικότητας. Κάνει πολύ περισσότερα όμως. Όταν μιλάμε για κινητικότητα, και αυτό ήδη προελέχθη, δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό σκοπός, απλώς είναι ένα μέσον για τα ανώτατα ιδρύματα να ανοίξουν τις πύλες τους στο διεθνή χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Το έρασμο συν, ως προς την κινητικότητα, ε, δεν προωθούμε τους επιστήμονες, αλλά και το προσωπικό ε, δεν το αναφέρατε, αλλά ε, εν υπάρχει στην έκθεσή σας, γιατί το διδακτικό προσωπικό, αν δεν ζήσει την κινητικότητα, δεν μπορεί να την προωθήσει στους φοιτητές. Γι' αυτό χαίρομαι, διότι φέτος με τον Erasmus ΣΥΝ θα προβούμε στην κινητικότητα 30.000 ε, διδασκόντων και φοιτητών εκτός Ευρώπης και υπάρχει κινητικότητα προς τα μέσα και προς τα έξω. Θα πρέπει να δείξουμε ότι και το ε, δικό μας προσωπικό και οι φοιτητές ε, θέλουν να κινούνται εκτός των συνηθισμένων ε, προορισμών, γιατί συνήθως προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο, στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε και εκτός Ευρώπης. Η κινητικότητα ε, αφορά και τη διεθνοποίηση, η οποία θα πρέπει να είναι πιο ε, συνεκτική, να προωθήσει κοινά προγράμματα που το κάνουμε και με το Erasmus Mundus και το Erasmus Sin και μέσα στα πλαίσια των ε, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι δελεαστικός προορισμός, αλλά θα πρέπει με συνεργασία και με ανταγωνισμό να προωθηθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και με το Erasmus Συν προσπαθούμε να ε, αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες και να προωθήσουμε την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το θέμα της ισότητας είναι ύψη της ε, σημασίας στο Erasmus Συν. Γι' αυτό τονίζουμε το θέμα της επιλογής φοιτητών που προέρχονται από ένα πιο ευάλωτο, ε, από μια πιο ευάλωτη κοινωνική προέλευση. Αυτό μας απασχολεί σύντητα, γι' αυτό ε, προωθούμε την ε, κινητικότητα των credits, γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν οι φοιτητές έρθουν στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό credits. Γιατί όταν αποκτούν ένα ευρωπαϊκό πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο υπάρχει η τάση να παραμείνουν στην Ευρώπη. Το έρασμο συν δεν είναι το μόνο μέσο που έχουμε για την διεθνοποιημένη στρατηγική. Έχουμε ε, διαλόγους πολιτικής με την Κίνα, την Ινδία και ε, το Μεξικό, Βραζιλία και άλλες χώρες προτεραιότητας και περιφερειακό πολιτικό διάλογο με τις ε, χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιής Μεσογείου και μιλάμε για το θέμα της αναγνώρισης των βαθμών αλλά και των διπλωμάτων. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων στη διάθεσή μας. Αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να διαβάσετε και αυτή την ανακοίνωση που εκδόθηκε δύο χρόνια πριν και η οποία είναι επίκαιρη ακόμα όταν ακούω ιδιαίτερα τα ευρήματα της εισήγησής σας. Οι απόφοιτοι φοιτητές, οι απόφοιτοι είναι ένα στοιχείο διεθνοποίησης και αυτό το βλέπουμε σε πανεπιστήμια και στην Ευρώπη. Ε, ενισχύουμε αυτά τα δίκτυα αποφύτων και είναι η καλύτερη πρέσβη μας, Υπάρχουν εθνικές στρατηγικές για την διεθνοποίηση και έχουμε και μία ευρωπαϊκή στρατηγική διεθνοποίησης που θα πρέπει να σχετίζεται με άλλες ε, εθνικές στρατηγικές, δηλαδή τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης και μετανάστευσης γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει η τάση να καταστήσουμε την Ευρώπη δελεαστική για σπουδές. Αλλά όταν οι φοιτητές δεν λαμβάνουν εύκολα θεωρήσεις, τότε αυτό οδηγεί σε ένα ε, αντίθετο, σε, στα αντίθετα αποτελέσματα, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις. Σας ε, δίνω την τελευταία λέξη. Έχετε την τελευταία λέξη. Ναι, η στρατηγική σας έχει συμπεριληφθεί στη δικιά μας τη μελέτη. Και ο συνάδελφος ε, το πόσο ξέρετε, συμμετείχε στην ομάδα η οποία εκπώνησε αυτή τη στρατηγική. Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν. <clears throat> Δεν έχω χρόνο βέβαια εδώ να σας πω πόσο το ευρωπαϊκό μοντέλο το ζηλεύουν και πολλοί προσπαθούν να το αντιγράψουν. Η Ευρώπη είναι πολύ τυχερή που μέσα σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, που υπάρχει διεθνοποίηση και στον τρόπο με τον οποίο κερδίζει κανείς το ψωμί του, ναι, υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, αλλά η συνεργασία είναι μέσα στο DNA της διεθνοποίησης. Το ευρωπαϊκό μας μοντέλο και τα όσα προσφέρουν τα προγράμματα Εράσμους και άλλα είναι στοιχείο κλειδί. Στο χρόνο που είχα ίσως δεν μπόρεσα να υπογραμμίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει και το προσωπικό. Δηλαδή, αν θέλουμε διεθνοποίηση των, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρειαζόμαστε και το προσωπικό, γιατί μπορείτε να φτιάξετε στρατηγικέ, μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε, αλλά οι ακαδημαϊκοί πρέπει να συμμετέχουν, να ενστερνίζονται όλη αυτή την προσπάθεια. Συνεπώ χρειάζεται η βοήθεια και των διοικητικών και όλων για να συνεισφέρουν. Δεν μπορείς να μάθεις μέσα σε μια τάξη για παράδειγμα, αν δεν έχεις βρει, που θα μένεις. Δεν μπορείς να σκεφτείς το μέλλον σου, αν σκέφτεσαι πώς θα έχεις τα χαρτιά για να είσαι εντάξει εκεί που μένεις. Τις άδειες παραμονής κλπ. Επιμένω πάντως, η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στην τάξη. Είναι σχέση ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο. Ναι στις στρατηγικές κλπ. Αλλά αν οι καθημαϊκοί δεν συμμετέχουν, δεν θα γίνει. Και βλέπουμε να υπάρχει στην Ευρώπη μια τάση. Το Ενωμένο Βασίλειο τελευταία εξέδωσε κάτι για την διδασκαλία και την εκμάθηση. Φυσικά ο ανταγωνισμός μας αναγκάζει να κοιτάμε τα αποτελέσματα της έρευνας πολύ. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι καθημαϊκοί πρέπει να πληρώνονται αρκετά για να μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν στην καλή εκπαιδευτική εμπειρία. Και το τελευταίο μου. Πιστεύω στην ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά πιστεύω και ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνοχή, να χρησιμοποιούμε τις ενέργειες. Όταν μιλάμε για κινητικότητα, εταιρικέ σχέσεις, διεθνοποίηση, ψηφιακή γνώση, όλα αυτά πρέπει να τα συγκεντρώσουμε σε ένα προϊόν. Θέλουμε να υπάρχει ένα διεθνοποιημένο πρόγραμμα μέσα σε έναν ψηφιακό χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκρος ενδιαφέρον το πρωινό ε, και η απάντησή σας αποσαφήνει σε ορισμένα πράγματα. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, θα πρέπει να δούμε την θετική ανταγωνιστικότητα με την προσφορά των πανεπιστημίων και την συνεργασία που είναι μια βασική αξία αλλά και πρόκληση για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα προσθήσουμε και στο μέλλον, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και στο μέλλον. Συγχαρητήρια για την εργασία σας και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τώρα, ένα λεπτό να συνοδεύσω την κυρία. Allora, Scusate, vorrei solo dirvi che concludiamo la nostra eh, riunione. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 ε, Δεκεμβρίου θα ε, ξανασυναντηθούμε, θα έχουμε τη διακυβερνητική συνέλευση. Θα ήθελα να είσαστε παρόντες, να το εξασφαλίσουν και οι επικεφαλείς ε, αντιπροσωπιών. Ευχαριστούν, ευχαριστώ και τους διερμήνες, σας ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να αποχωρήσετε από την αίθουσα γιατί θα συνεδριάσουν οι συντονιστές